Uh, Ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε σε αυτή τη δημόσια ακρόαση, κοινή δημόσια ακρόαση των Επιτροπών Απασχόληση και Διεθνού Εμπορίου για την απασχόληση και τι κοινωνικέ πτυχέ τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων. TTIP. Θα πω λίγα λόγια στη δική μου γλώσσα, τα σουηδικά, και μετά θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο τη Επιτροπή ΣΥΝΤΑ. Έχουμε, ε, τρέφουμε σοβαρές ελπίδες για τη Συμφωνία Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης συνελεγών και Επενδύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πολιτειών. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και σοβαρές ανησυχίες. Αναφέρονται τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, το περιβάλλον, η ανάπτυξη και η εξελίξη στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε τι ε, προτεραιότητες υπάρχουν στην Ευρώπη της κρίσης, όπως ε, έχει δημορφωθεί αυτή τη στιγμή, και κάποιες πτυχές προσπαθούμε να τις καλύψουμε μέσω της ε, συμφωνίας αυτής, όμως φοβόμαστε ότι θα επιβαρυνθούν άλλοι τομείς. Σε αυτή τη στιγμή που υπάρχει εκτεταμένη ενεργεία στην Ευρώπη, πρέπει κάτι να κάνουμε καθήκον μας ως μελών του Κοινοβουλίου και επειδή μπορούμε σε ένα βαθμό να επηρεάσουμε από τη συμφωνία, θα πρέπει να μελετήσουμε καλά τις λεπτομέρειες, όλα τα ζητήματα και να δούμε τι θα μπορούσε να συμβεί και να προσπαθήσουμε να θέσουμε σαφείς στόχους, να δούμε τι ακριβώ θέλουμε να πετύχουμε. Γι' αυτό είναι πολύ καλό ε, να έχουμε αυτή την κοινή συζήτηση, ώστε να διατρέξουμε κάποια από τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν με τις ενδιαφερόμενες επιτροπές. Να δώσω τώρα το λόγο στον Μπεντ Λάγκε, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Ευχαριστώ, Νίτο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, πράγματι, το ζήτημα των επιπτώσεων στην απασχόληση και στα κοινωνικά πρόταπα και πώς αυτά θα επηρεαστούν από μια συμφωνία ελεύθερου εμπειρίου είναι θεμελιώδες για την αξιολόγηση μιας τέτοιας συμφωνίας. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι αν ε, θεσπιστούν σωστά οι όροι, μπορεί να ενισχυθεί η απασχόληση στην Ευρώπη και μπορεί να συμβάλλει μια τέτοια συμφωνία στο να βελτιωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αλλά αυτό εξαρτάται από τους όρους της συμφωνίας. Και νομίζω ότι σε αυτό θα επικεντρωθούμε σήμερα στη συζήτησή μας. Στο πώς θα καταφέρουμε να δημορφώσουμε τους όρους αυτής της συμφωνίας με τέτοιον τρόπο, ώστε να προκύψουν και βελτιώσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί είναι σαφές ότι μια εμπορική συμφωνία μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον πληθυσμό, από τους λαούς μόνο εφόσον υπάρχει νομοθεσία που θα διασφαλίζουν τους κανόνες εργασίας. Και από αυτή την άποψη μια σύγχρονη συμφωνία εμπορίου δεν θα πρέπει να περιστρέφεται μόνο γύρω από τη μείωση των δασμών, αλλά θα πρέπει να έχει στο επίκεντρό της και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και αν κανείς εξετάσει το TTIP, Ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων στη ΣΥΠΑ υπάρχουν κάποιες προκλήσεις. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν 8 συμβάσεις, βασικές συμβάσεις για τα... Ε, συμβάσεις για την, ε, για, την εργασία. Μόνο δύο από αυτές οι ΙΠΑ έχουν κυρώσει. Ενώ τις άλλες έξι όχι. Τα τελευταία χρόνια στις συμφωνίες εμπορίου πάντοτε κοιτάζουμε να υπάρχει και μια παράγραφος, ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Να γίνονται σεβαστές, σεβαστά τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Προσπαθούμε να βελτιώνουμε τους κανόνες και να εξασφαλίζουμε τη δεσμευτικότητα αυτών των διατάξεων και αυτών των βασικών κανόνων εργασίας και των βασικών περιβαλλοντικών προτύπων και βεβαίως με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει κανείς να εξετάζει και τις ε, επενδύσεις. Όταν μιλάμε σήμερα για τα ISDS, συνήθως η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την εξασφάλιση των επενδυτών, αλλά Σχεδόν ποτέ η συζήτηση δεν περιστρέφεται για το αν οι επενδυτέ αυτοί θα πρέπει να καταβάλουν και ορισμένε προσπάθειε για τα δικαιώματα των εργαζομένων ή για το περιβάλλον. Εμείς λοιπόν θέλουμε να αναπτυχθεί περαιτέρω η εταιρική κοινωνική ευθύνη και θέλουμε επίσης η κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει ενεργότερα στην ε, εφαρμογή αυτών των κοινωνικών προτύπων Και γι' αυτό νομίζω ότι και ο ρόλος των συμβουλευτικών επιτροπών των εργαζομένων θα είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια γκάμα ερωτημάτων και ζητημάτων που θα πρέπει να απαντηθούν αν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια καλή εμπορική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και από αυτή την άποψη ανυπομονώ να ακούσω τι έχει να μας πει η Κομισιόν πως εκείνη ε, αξιολογούν τις διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για τα εργασιακά δικαιώματα και το περιβάλλον και χαίρομαι που είναι εδώ και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ο κ. Μπερσέρο αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι είναι εκπρόσωπος εδώ και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας η οποία πρόσφατα εξέδωσε και μια μελέτη στην οποία αναλύονται διάφορες ε, εμπορικές συμφωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο και έτσι νομίζω ότι μπορούμε να σχηματίσουμε και μια εικόνα για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί μια καλή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Μπέντ Λάγκε. Να καλωσορίσω τον κύριο Ιγνάφιο Γκαρθία Μπερθέρο, τον επικεφαλής διαπραγματευτή ε, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα του δώσω το λόγο για να μας κάνει μια εισαγωγή. Ευχαριστώ. Είναι τεράστια χαρά να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας την συμφωνία TTIP ε, από την σκοπιά του αντικτύπου που θα έχει στην απασχόληση και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Στην ε, αρχική μου αυτή εισήγηση θα ήθελα να επικεντρωθώ όχι μόνο στο κεφάλαιο των εργασιακών ζητημάτων του TTIP, γιατί θα είναι ένα σημαντικότατο σκέλος της συζήτησης, αλλά επίσης να δούμε σφαιρικότερα το πώς η συμφωνία TTIP θα επηρεάσει όσα αφορούν την απασχόληση και τις ε, συνθήκες των κοινωνικών δικαιωμάτων. Πιστεύουμε ότι η συμφωνία που διαπραγματευόμαστε με τη ΣΥΠΑ είναι φιλόδοξη και θα φέρει πραγματικές βελτιώσεις ως προς την πρόσβαση στην αγορά Πιστεύουμε ότι ο αντίκτυπος θα είναι θετικός και για τις δουλειές και για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν εξαιτία της συμφωνίας αυτής, όμως αυτό που μπορεί κανείς να πει με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας είναι ότι πολλές ε, θέσεις εργασίας στην Ευρώπη εξαρτώνται από το διατλαντικό εμπόριο. Περίπου 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτώνται από το εμπόριο αυτό. Όσο λοιπόν πετύχουμε να διευρύνουμε και να αντίνουμε το διατλαντικό εμπόριο, τόσο θα συμβάλλουμε προς την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία που να είναι και φιλόδοξη αλλά και ισορροπημένη. Δεν θέλω να περάσω σε υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες στα πλαίσια αυτής της αρχικής εισήγησης, απλώς να σας δώσω κάποια σημαντικά στοιχεία ως προς την πρόσβαση στην αγορά, τους δασμούς, τις υπηρεσίες και τις δημόσιες προμήθειες. Έχουμε πρόσφατα συνάψει μια φιλόδοξη συμφωνία με τον Καναδά, η οποία μας δίνει κάποιους βασικούς δείκτες για το τι ύψος φιλοδοξιών μπορούμε να επιδιώξουμε στις διαπραγματεύσεις μας με τη ΣΥΠΑ εξαλείψαμε περίπου το 99% των δασμών στη συμφωνία μας με τον Καναδά, ενώ παράλληλα διατηρήσαμε την προστασία για κάποιους από τους πιο ε, ευαίσθητους και ευάλωτους τομείς της ε, οικονομίας μας καταφέραμε να έχουμε μια φιλόδοξη συμφωνία για τις υπηρεσίες βάσει ενός αρνητικού καταλόγου αλλά προστατεύοντας τις δημόσιες υπηρεσίες και χωρίς να αναλάβουμε καμία δέσμευση για τον οπτικοακουστικό τομέα. Εδώ λοιπόν να είμαι σαφής. Η προσέγγιση μας για τις δημόσιες προμήθειες είναι πρώτον ότι δεν θα αναλάβουμε δεσμεύσεις και δύο ότι θα διαφυλάξουμε πλήρως τα δικαιώματα των κυβερνήσεων να αποφασίζουν. Να αποφασίζουν κατά πόσον κάποιες υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από τον δημόσιο τομέα. Αυτή είναι η προσέγγιση που έχουμε ως τώρα σε όλες τις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις και αυτή την προσέγγιση θα διατηρήσουμε και στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Επίσης, πετύχαμε σημαντικά αποτελέσματα σε δύο τομείς που θα είναι δυσχερείς ε, και θα μας δυσκολέψουν στις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Όμως, εκεί έχουμε πολλά βασικά συμφέροντα. Τη μη διακριτική μεταχείριση στις δημόσιες προμήθειες και την ε, προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει τη συμφωνία TTIP είναι ότι στι δημοτέ αυτέ προσπαθούμε να επιτελέσουμε πρόοδο και ω προ την μεγαλύτερη συμβατότητα των ρυθμίσεων των ΗΠΑ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, ό,τι κάνουμε ε, στο επίπεδο των ρυθμιστικό βασίζεται σε δύο βασικέ αρχέ. Πρώτον, δεν ε, ε, υποβαθμίζουμε το επίπεδο προστασία μα, σε καμία περίπτωση δεν διακυβεύουμε την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, του περιβάλλοντο και τη υγεία στο πλαίσιο μια εμπορική συμφωνία και επιπλέον διατηρούμε πλήρω τη ρυθμιστική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ε, έγκριση νέων κανόνων. Με αυτά τα αρχικά σημεία εφετηρία, πιστεύουμε ότι μπορούν να είναι σοβαρότατα τα πλεονεκτήματα από αυτή τη συμφωνία για την απασχόληση και τι θέσει εργασία. Και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε σημαντικότητα αποτελέσματα και στον τομέα το ρυθμιστικό. Να σα δώσω απλώ δύο παραδείγματα. Το εμπόριο το ε, ε, εμπόριο τη αυτοκινητοβιομηχανία είναι πολύ σημαντικό μέρο των εξαγωγών προ τι ΗΠΑ και πιστεύουμε ότι η συμφωνία αυτή θα αυξηθούν ακριβώ οι εξαγωγέ. Βεβαίω είναι πολύ σημαντικό ότι οι δασμοί είναι 2,5% μόλι για το εμπόριο αυτό στι ΗΠΑ, αλλά υπάρχουν και κανονισμοί ασφαλεία και προστασία που έχουν εξαιρετική σημασία για την αυτοκινητοβιομηχανία. Οπότε το να πετύχουμε ε, καλύτερα αποτελέσματα ω προ τι εξαγωγέ αυτοκινήτων προ τι ΗΠΑ, όλο αυτό θα δείξει γενικότερα πώς θα πετύχουμε μεγαλύτερη ρυθμιστική ε, συμβατότητα για την προστασία. Το ίδιο και με ε, τα, με τα όρια που έχουμε για, τις, για τους ελέγχους, την γραφειοκρατική σκοπιά. Θα πρέπει η επικάλυψη ελέγχων ή επιθωρήσεων που κάποιες φορές απαιτούνται και από την πλευρά των Αμερικανικών αρχών να εξελιχθούν. Αυτό θα είναι ένα σημαντικότατο βήμα για να αυξηθούν πάλι οι εξαγωγές μας. Και αυτό τα αξιοποιούμε σε τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία, τα ιατρικά ε, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και βεβαίως ε, και για άλλους τομείς. Όπως είπε και ο Μπεν Πλάνγκε, από την ε, συμφωνία μας με την Κορέα και μετά βλέπουμε ότι όλες οι πρόσφατες συμφωνίες μας συμπεριλαμβάνουν ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνει και ένα κεφάλαιο για την ε, αγορά εργασίας και ένα άλλο για το περιβάλλον. Στην περίπτωση των ΗΠΑ είναι σημαντικό ότι ήδη έχει συμβεί και πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για, την, για τα εργατικά και την, το περιβάλλον Έχει συμβεί να έχουμε ήδη κάποιε σχετικέ διαπραγματεύσει. Από όλε τι χώρε λοιπόν με τι οποίε διαπραγματευτήκαμε, ίσω είναι η μόνη περίπτωση που και οι δύο ξεκινήσαμε από το βασικό ε, αρχικό ε, σημείο ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, προστασία των εργατικών δικαιωμάτων. Φυσικά υπάρχουν διαφορέ μεταξύ του αμερικανικού και του ευρωπαϊκού μοντέλου και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε σε αυτέ τι διαπραγματεύσει είναι να δούμε πώ θα συμβιβάσουμε τι διαφορέ μα. Όχι βάσει του ελάχιστου κοινού παρανομαστή, αλλά προσπαθώντα να φέρουμε πραγματικέ βελτιώσει ω προ το τι θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα κεφάλαια αυτά. Το εφαλτήριο για τα θέματα αυτά είναι το κεφάλαιο που διαπραγματευτήκαμε σχετικά με τον Καναδά και ήταν πολύ επιτυχημένο. Βεβαίω, καλό θα ήταν όλοι να έχετε δει το κεφάλαιο που συμπεριλάβαμε στη συμφωνία μα με τον Καναδά για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με στοιχεία για τα εργατικά δικαιώματα και το περιβάλλον. Αυτά είναι διαθέσιμα στον τόπο μα. Και πολύ σημαντικό θα ήταν να ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή και στι διαπραγματεύσει με τη ΣΥΠΑ. Όμω, σε κάποιου τομεί μπορεί να πάμε και παραπέρα σε όσα θα συμφωνήσουμε με τη ΣΥΠΑ σε σχέση με τον Καναδά. Χαίρομαι πολύ που υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι του ILO, διότι θέλω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για το όλο ζήτημα αλλά κάτι που ανέκαθεν ήταν πολύ σημαντικό για μας σε όλες τις εμπορικές μας συμφωνίες ήταν να έχουμε παραπομπές στον, στο, διεθνή, στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και να λαμβάνουμε υπόψη τα πρότυπα που ε, προβλέπει ο ILO. Εδώ λοιπόν αυτό το κάναμε και στη συμφωνία με τον Καναδά και στην ε, τι δημοτεύσει αυτέ, ασχέτω με το αν έχουν κυρωθεί ή όχι οι συμβάσει του ΕΛΟ, ε, φροντίζουμε να δεσμευόμαστε ότι η εγχώρια νομοθεσία μα συνάδει με τι αρχέ και όσα προβλέπει για τα δικαιώματα η κάθε, κάθε μια από αυτές τις συμβάσεις. Έπειτα, στην περίπτωση του Καναδά, πήγαμε παραπέρα από τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε σχέση με τις προτεραιότητες για την εξωπρεπή εργασία του ΑΕΛΟ και άλλες πτυχές των εργατικών δικαιωμάτων, όπως τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας και σε όλες τις συμφωνίες μας θα συνεχίσουμε, όπω όλε μα τι συμφωνίε μα μάλλον, θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε διαρκεί προσπάθειε για την κύρωση των συμβάσεων του ΑΕΛΟ που δεν έχουν ακόμη κυρωθεί. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο των συμφωνιών μα είναι ο ρόλο τη κοινωνία των πολιτών. Στη συμφωνία με τον Καναδά έχουμε θεσπίσει ένα σύστημα όπου και οι δύο πλευρές μιας συμφωνίας έχουν ε, συμβουλευτικά σώματα με μέλη από την κοινωνία των πολιτών για τα εργατικά και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και ένα φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών με αναγνωρισμένο ρόλο ε, παρακολούθησης των διαπραγματεύσεων σε αυτά τα δύο κεφάλαια. Αυτό κάναμε στις διαπραγματεύσεις μας με τον Καναδά και νομίζω ότι αν τα κοιτάξετε θα δείτε ότι το επίπεδο λεπτομεριών είναι πολύ σημαντικό. Εδώ νομίζω οι συμφωνίες μας μπορούν να πάνε παραπέρα στην περίπτωση των ΗΠΑ ε, και τη συμφωνία μα με τον ΗΠΑ ω προ την κοινωνία των πολιτών και τη διαδικασία παρακολούθηση. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο νομίζω πρέπει να σκεφτούμε είναι πόσο πολύ μπορεί να αναπτυχθεί ο ρόλο τη κοινωνία των πολιτών και αν πρέπει να περιοριστεί στην βιώσιμη ανάπτυξη και το κεφάλαιό τη ή αν πρέπει να διευρυνθεί στη συμφωνία TTIP. Είναι σαφέ ότι είναι πολλέ οι πτυχέ που μπορούμε να διαπραγματευτούμε στο πλαίσιο τη συμφωνία TTIP και που θα ενδιαφέρουν και του κοινωνικού μα εταίρου. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, από τα ζητήματα που μας απασχολεί είναι στο ρυθμιστικό επίπεδο πώς να βεβαιωθούμε ότι στο μέλλον οι θεσμοί θα διευκολύνουν τη ρυθμιστική συνεργασία. Ένα από τα στοιχεία που θα ήθελα να εξετάσουμε σε αυτό το πλαίσιο είναι πώς οι διαφορετικές συνιστώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι επιχειρήσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει παίζουν ένα ρόλο στην όλη αυτή ε, αλληλεπίδραση μέχρι να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και ρυθμιστική συνεργασία. Ω προ το που έχουμε φτάσει στι διαπραγματεύσει, είχαμε εντατικότατε συζητήσει με τη ΣΥΠΑ τον τελευταίο χρόνο και τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορέσουμε να υποβάλουμε πριν τον επόμενο διαπραγματευτικό γύρο μια συγκεκριμένη πρόταση για το κεφάλαιο αυτό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και όπως ξέρετε, μόλις η πρόταση αυτή υποβληθεί, στις ΗΠΑ θα δημοσιευτεί και όπως ανακοίνωσε η Επίτροπος Μάλστρομ θα είναι κάτι που θα μπορείτε να το ε, δείτε κι εσείς. Δηλαδή μόλις ε, ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο σε επίπεδο κρατών μελών και με το Κοινοβούλιο θα δημοσιευτούν όλα στον ιστοτοπό μας. Μπορούμε όμως ήδη να δούμε κάποιες λεπτομέρειες των στοιχείων που μάλλον θα συμπεριληφθούν στην γραπτή μας πρόταση. Ευχαριστώ. Κύριε Μπεσέρο, σας ευχαριστούμε. Και τώρα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κόρλια Κουλιμπαλία του Διεθνούς Γραφείου εργασία, της Διευθύνσεως Ερευνών. Έχετε και κάποιες διαφάνειες. Ναι, ναι, έχω μια διαφάνεια PowerPoint. Να σας ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα για την πρόσκλησή σας Είμαι ανώτερη υπάλληλο, οικονομολόγο του Διεθνούς Γραφείου Έχουμε μια ομάδα για την παγκοσμιοποίηση και τα, τους κανόνες, <clears throat> τα στάνταρ για την απασχόληση και έχουμε εδώ πέρα ένα πολιτέ πρόγραμμα το οποίο αφορά την αποτελεσματικότητα των εργασιακών διατάξεων σε αυτές τις ε, συμφωνίες και πρόσφατα έχουμε δημοσίευσει μια έρευνα όσον αφορά αυτέ τι ε, εμπορικέ συμφωνίε. Έχω κάποια έγραφα θα δώσω. Ε, υπάρχουν στο, στην αίθουσα στην είσοδο. Να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτές τις ε, διατάξεις, τις ε, εμπορικέ συμφωνίες, τι γίνεται από πλευράς θεσμικής και έχουμε και κάποιες συγκεκριμένες μελέτες και επίσης κάποιες συστάσεις. Και να δούμε τώρα ποιος είναι ο ρόλος της σε σχέση με αυτές τις διατάξεις που αφορούν τις απασχολήσεις και αυτό αφορά τι άριστε ε, πρακτικών με Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΠΑ, αλλά έχουμε και άλλα παραδείγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε ε, αυτού του είδου ε, την διαδικασία του TTIP και δεν έχουμε κάνει τέτοια ανάλυση, γιατί η ανάλυση μα εστιάζεται σε αυτού του είδου τι συμφωνίε, αυτέ που έχουν ήδη κυρωθεί. Οπότε, θα σα το προσθέσω εξή στον χρόνο που έχω πρώτα πρώτα μια γενική άποψη του πού βρισκόμαστε όσον αφορά τον πολλαπλασιασμό αυτών των διατάξεων για την απασχόληση σε εμπορικέ διατάξει. Θα σα πω ποιο είναι ο ρόλο του Διεθνού Γραφείου Εργασία σε σχέση με τα <clears throat> πρότυπα. Επίση θα πρέπει να δούμε τα κοινά σημεία ε, για τι προσεγγίσει Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΠΑ. Και να δούμε επίση τι μπορεί να κάνει ε, στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Εδώ, μπορεί να δείτε εδώ ε, αθρηστικά τον αριθμό των ε, συμφωνιών μεταξύ 1990 και 2014. Από τότε που έχουμε τέτοιου είδους διατάξεις για την απασχόληση ε, από το 1994 βλέπετε ότι αυξάνεται ο αριθμός και φτάνουμε στις 68 σε 68 εμπορικές συμφωνίες που έχουν διατάξεις απασχόλησης το 2014. Είναι το σύνολο. Δύσκολο να διακρίνετε τώρα αυτά τα οποία αναγράφονται σε αυτό το διάγραμμα, αλλά εδώ πέρα λέει τι έγινε από το 2010 και δείχνει τον αριθμό των συμφωνιών διατάξεις απασχόλησης που ετέθησαν σε εφαρμογή το 2010 σαν ποσοστό του συνόλου των εμπορικών συμφωνιών. Συνολικά έχουμε 28 συμφωνίες με διατάξεις απασχόλησης από το 2010. Το 1 τέταρτον προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την εξαίρεση του 2012 το ποσοστό των συμφωνιών αυτών με τέτοιες διατάξεις βαίνει αυξανόμενο αυτό λόγω του ότι έχουν συναυθεί συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΙΠΑ και Καναδά γιατί εκεί υπάρχει μια παράδοση να έχουμε τέτοιες διατάξεις σε αυτές τις συμφωνίες αλλά επίσης και την νέων εμπλεκομένων, Κορέα, ΕΦΤΑ ε, και άλλες συμφωνίες συνεργασίας με Κίνα και Χιλή. Εδώ βλέπετε επίσης μια άποψη αυτών των ε, συμφωνιών. Έχουν εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη ΣΥΠΑ οι χώρες οι μπλε και έχουν τέτοιες διατάξεις στις ε, συμφωνίες. Ε, πράσινο, πράσινο είναι οι χώρες που δεν έχουν ε, συνάψει συμφωνίες τέτοιες. Και εδώ βλέπετε και επίσης υπάρχουν και κάποιες που δεν έχουν τέτοιες συμφωνίες με Ευρωπαϊκή Ένωση ή είπα τώρα βλέπουμε επομένως ότι έχουμε πολλαπλασιασμό τέτοιων διατάξεων στις ε, εμπορικές συμφωνίες και αυτό έχει συμβεί όχι μόνο σε Ευρωπαϊκή Ένωση και είπα, αλλά και παγκοσμίω. Για να δούμε τώρα ποιο είναι ο ρόλο του Διεθνού Γραφείου Εργασία, ιδίω όσον αφορά τα πρότυπα απασχόληση. Η εντολή του ILO είναι να ε, ε, φτιάχνει τέτοια πρότυπα και να βροντίζει για την ε, κύρωση και εφαρμογή τους. Όλα αυτά γίνονται σε σχέση με τα εμπορικές συμφωνίες και σε 60% των περιπτώσεων όταν έχουμε μία παραπομπή σε τέτοιες διατάξεις και σε τέτοια πρότυπα αναφερόμαστε στην διακήρυξη του 98 του ΕΛΟ όσον αφορά τα δικαιώματα στην εργασία ή στις βασικές συνθήκες που διέμουν τον ΕΛΟ. Επομένω έτσι υπάρχει μια εντολή ούτως ώστε να προάγεται η κύρωση και η υλοποίηση αυτών και αυτό πρέπει να το κάνουν τα κράτη-μέλη. Και επίση υπάρχει και ένα εποπτικό μηχανισμό. Και έτσι οι επιτροπέ του ΑΕΛΟ μπορούν να έχουν κάποιε εκθέσει όσον αφορά τη συμμόρφωση για τα πρότυπα αυτά. Γίνονται κατά διαστήματα και έτσι αυτό είναι ένα εργαλείο εποπτεία. Για να δούμε τώρα πώς εμπλέκεται ο ΑΕΛΟ όσον αφορά το τι γίνονται αυτά τα διεθνή στάνταρ απασχόληση αφού έχουν ενσωματωθεί στις εμπορικέ συμφωνίε. Έχουμε τεχνική συνεργασία που διευκολύνει την ε, εφαρμογή αυτών των ε, προτύπων. Και επίσης έτσι αξιολογείται ε, το, το αν αυτά έχουν ενσωματωθεί στις εμπορικέ συμφωνίε. Να έχουμε εδώ πέρα τρία παραδείγματα συμφωνιών. ΙΠΑ, Κολομβία, στο, πρόγραμμα δράση και, τα τρία παραδείγματα έχουν να κάνουν με τη ΣΥΠΑ, αλλά εδώ σας δείχνει τι έκανε ο ILO στις χώρες που συνέπηξαν αυτές τις συμφωνίες, ε, είτε με δημιουργία παραγωγικών δυνατοτήτων, ε, με επιθεωρήσεις, με εποπτεία, σε όλα τα επίπεδα ή με κάποια διαδικασία τριμερή. Τώρα θα σας τονίσω μια συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά την ε, συμφωνία, την εμπορική, είπα, Καμπότζης, γιατί πιέζει ο χρόνος. Και ε, αυτό αφορά την συμφωνία κλώστου εφαντουργικά του 1999 με τις είπα είναι πλάκη σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την ρύθμιση ο ILO. Είχαμε κάποιους ε, δείκτες για αξιολόγηση της συμμόρφωσης για το τι γίνεται με τις εξαγωγές, τα σχετικά εργοστάσια, αυτού του τα πρότυπα και επόπτευσε την εφαρμογή αυτών των προτύπων. Επίσης, παρακολουθήσαμε την εφαρμογή και είχαμε κάποιες εκθέσεις για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα. Υπήρχαν, αλλά βεβαίως τα βελτιώσαμε. Και μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο στο website του Γραφείου εργασία. Επίσης, αν δείτε μια ματιά στους εποπτικούς μηχανισμούς, θα δείτε ότι, ότι πρώτα-πρώτα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ε, τη βοήθεια αυτών των της ΕΠΑ και των Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης στα πλαίσια των συμφωνίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, και αυτό το χρησιμοποίησαμε ως σημείο αναφοράς στον υπόλοιπο χρόνο τώρα για να δούμε τι γίνεται με την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα στις πιο πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες για κάποια βασικά σημεία όπως η παραπομπή ε, στα διεθνή πρότυπα για την συνεργασία, εποπτεία και επίλυση διαφορών. Ακόμα δεν έχουμε περιλαβεί εδώ τη συμφωνία με τον Καναδά γιατί ακόμα δεν έχει κυρωθεί. Τώρα, για την παραπομπή σε αυτά τα διεθνή πρότυπα όλα τα μέλη του ILO δεσμεύονται, όπως σας ανέφερα, σύμφωνα με την διακήρυξη του 98 και βλέπουμε και από την Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΥΠΑ, ΕΕ, έτσι βελτιώνονται και τα διεθνή πρότυπα η Ευρωπαϊκή Ένωση όλες τις ε, συμβάσεις και συμφωνίες τις έχει κυρώσει και αυτό οδηγεί σε αποτελεσματική εφαρμογή. Ας πούμε την συμφωνία με την Κορέα, τονίζουμε το ότι θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες κύρωσης και επίσης ε, έχουμε την συμφωνία με την ε, Κεντρική Αμερική που και αυτή έρχεται να παραπέμψει στις ε, συμφωνίες της, του Εθνικού Εργασίας. Επίσης ε, με τις, με τις έχουμε την ε, υλοποίηση, εφαρμογή εθνικών νομοθεσιών. Και εδώ είχαμε μεταρρυθμίσεις στην νομοθεσία πριν την κύρωση. Και αυτό γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Με στο Μεξικό και για άλλες συμφωνίες, οπότε αυτές οι μεταρρυθμίσεις ήταν κέρδος για τους εργαζομένους μπήκαν σε συνδικάτα και επίσης μπήκε τέλος σε κάποιες δυσμενείς διακρίσεις. Όσον αφορά τώρα την εποπτεία και συνεργασία, η πρόεδρος. used your time. Έχετε εξαντλήσει το χρόνο σας. Μας μπορείτε να κλείσετε το, θέμα της επίλυσης των θα είναι πάρα πολύ βασικό στον τη διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω μια διαδικασία ε, διαβούλευση με ε, κάποιους κυβερνητικού του κυβερνητικούς και υπάρχει, υπάρχουν δεσμευτικές αποφάσεις και υπάρχει παραπομπή στον ρόλο του ILO ε, που συμβουλεύει και εμπλέκεται γιατί σας είπα υπάρχει κάτι παραπάνω διότι εκεί πέρα οι διαβουλεύσεις για τα εργατικά περνούν από κάποια συνεργατική συμφωνία και μπορούν να οδηγήσουν και σε κυρώσεις μόνο, μόνο μία περίπτωση θα σε αυτή τώρα είναι η τωρινή υπόθεση που αφορά την Γουατεμάλα τώρα για να τονίσουμε ε, τι έγινε με την Γουατεμάλα και τον ρόλο του ΑΕΛΟ είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό για αυτό που συζητούμε είναι πάρα πολύ ε, πρόσφατη περίπτωση, πρώτη φορά που μια τέτοια υπόθεση απασχόλησης έφτασε σε επιδιαιτησία, ξεκίνησε τον Νοέμβριο μετά από έξι χρόνια της προκριτικής διαδικασίας, από το 2006 δηλαδή, και ο ρόλος ε, του Γραφείου Εργασίας είναι το ότι οι τούντες προέβαλαν σε επιχειρήματα τις παρατηρήσεις των ε, εποπτικών επιτροπών του ILO, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές εργασία κλπ. Και εδώ υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία όσον αφορά το τι έγινε ε, στην τη Γοτεμάλα και σε παλαιότερες ε, υποθέσεις για συγκεκριμένους στόχους, κάποιες ε, συστάσεις για τα εργασιακά δικαιώματα, για τη δημιουργία παραγωγικών δυνατήτων. Η Γοτεμάλα έχει ένα μήνα να απαντήσει, αλλά όμως συνεχίζουν οι ΙΠΑ να φροντίζουν για τα εργατικά δικαιώματα, τώρα για τον ρόλο του ΑΕΛΟ. Πέραν του παραδοσιακού ρόλου του Γραφείου Εργασία έχουμε και την εποπτεία για τα εργατικά πρότυπα, έχουμε τα θέματα της εφαρμογή και έχουμε και άλλους δύο τομείς που μπορεί να διαδραματίσει με πιο σημαντικό ρόλο ο ΑΕΛΟ σε σχέση και με ε, τις διάρκειες της TTIP. Έχουμε το θέμα της ε, συνέπειας με τα διάφορα μέσα ε, που χρησιμοποιεί ο ΕΛΟΣ στο έργο του και τον ε, μηχανισμό διαβούλευσης, αλλά όμως έχουμε στοιχεία από πρόσφατες ερεύνες που οδηγούν στο ότι έχουμε πιο ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σε αυτό το ρόλο του ILO και υπάρχουν συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με την άχρηση των θέσεων απασχόλησης αλλά πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη ανάλυση ε, ε, κυρίως για τα ποιοτικά στοιχεία των θέσεων απασχόλησης έχει ασχοληθεί το τμήμα ερεύνης μας και το 2015 πρόκειται να αποτελέσματα. Ο λόγος στον κύριο Τζένκις από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις δύο επιτροπές για το γεγονός ότι λάβαμε πρόσκληση ως Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων που εκπροσωπεί τι ομοσπονδίες, τα συνδικάτα σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα πέρα. Η συνομοσπονδία μας έχει θέση για το TTIP και έχουμε θέσει και κάποιες κόκκινες γραμμές. Το ένα είναι για το ISDS. Ξέρω ότι δεν θα θέλετε να το συζητήσουμε σήμερα αυτό. Υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την εξασφάλιση των δημοσίων υπηρεσιών και από αυτή την άποψη χαίρομαι που ο κ. Μπερσέρο αναφέρθηκε στους στόχους ε, της ε, Κομισιόν να εξασφαλιστούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει ένας αρνητικός κατάλογος. Ε, κάτι τέτοιο τουλάχιστον καταλήχθηκε στη συμφωνία με τον Καναδά, οπότε θα συνεχιστεί η συζήτηση. Αλλά αφού σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα, ας επικεντρωθούμε σε αυτά. Βασικά, εμείς θέλουμε έναν ε, ευρύτατο, ένα ευρύτατο κεφάλαιο για την εργασία. Προτού όμως περάσουμε σε αυτό, χαίρομαι που η εκπρόσωπος του ILO αναφέρθηκε στις ποιοτικέ διαστάσεις της έρευνας για τις θέσεις επασχόλησης. Εμείς είμαστε αβέβαιοι όσον αφορά την δημιουργία αξιοπρεπών ε, συνθήκων ε, απασχόλησης από το TTIP οι αρχικές ε, εκθέσεις αξιολόγησης στην οποία, στις οποίες η Κομισιόν ε, βάσισε τις προβλέψεις της ε, βασίστηκαν στην ε, γενική ισορροπία, στην αρχή της γενικής ισορροπίας και αυτό το μοντέλο το χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα και δεν νομίζω ότι η Παγκόσμια Τράπεζα είναι το πρότυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την ε, δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Αλλά ακόμη και εκείνη η έκθεση μιλούσε μόνο για 0,5% αύξηση του ΑΔΕΠ σε ε, ορίζοντα 10 ετών. Δεν μας είπα καθόλου τι είδου θέσει θέσεις θα ήταν αυτές και πρόσφατα το Πανεπιστήμιο ε, εξέδωσε μια μελέτη η οποία προβλέπει τα αντίθετα. Ότι θα υπάρξει απώλεια θέσεων απασχόλησης ε, λόγω του TTIP. Και η δική του μελέτη βασίζεται σε ένα διαφορετικό μεντέλο που το χρησιμοποιεί ε, το χρησιμοποιούν οι υπηρεσίε του ΟΗΕ. Αν λοιπόν το ζήτημα που συζητάμε είναι η θέσει απασχόλησης Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι πέρσι τον ε, Ιούλιο αναβλήθηκε η έκδοση της τεχνικής έκθεσης που επρόκειτο να δημοσιευθεί. Οπότε αναρωτιόμαστε τι έγινε με αυτήν. Εμείς δεν είμαστε καθόλου σίγουροι λοιπόν για το πού πάει το πράγμα σε σχέση με τις ε, θέσεις απασχόλησης. Δεν, δεν λέμε ότι σίγουρα θα χαθούν θέσεις απασχόλησης, αλλά δεν είμαστε καθόλου ε, ε βέβαιοι για την αύξησή τους. Θα χαθούν θέσεις απασχόλησης αυτό συμβαίνει πάντα σε αυτές τις ε, συμφωνίες. Σε κάποιο σημείο γίνεται αναφορά στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, αλλά η χρηματοδότηση αυτού του Ταμείου είναι εξαιρετικά περιορισμένη, το σύστημα είναι πραγματικά ακατανόητο και κάποιοι ε, θα ήθελαν ε, να το, να καταργηθεί και να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια αυτά για τη γεωργία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα χρειαστούμε κάποιο μηχανισμό προσαρμογής. Δεύτερον, για την ε, κανονιστική συνοχή. Όπως είπαμε το TTIP δεν αφορά μόνο την ε, πρόσβαση στην αγορά. Μπορεί να θυμάστε το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο βέβαια δεν ήταν ε, θέμα της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου αλλά της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και εκεί έγινε προσπάθεια να καθοριστούν ορισμένα πρότυπα και δεν έγινε ποτέ. Καταλαβαίνω ότι η, ρυθμιστική συνοχή θα πρέπει να είναι τμήμα μιας συμφωνίας αλλά εμένα το, το ερώτημα που με απασχολεί είναι τι ανταλλάγματα θα δοθούν στους εμπόρους όσον αφορά την ε, πρόσβαση στην αγορά. Εκεί που νομίζω ότι ο Ιγνάσιο έχει δίκιο είναι ότι αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να διαμορφωθεί και από τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό το, το Διατλαντικό Συμβούλιο είχε ε, συμβούλους από τους κοινωνικούς εταίρους αλλά στην παρούσα διαδικασία η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και ο αντίστοιχος φορέας από τη ΣΥΠΑ αποκλείστηκαν από τις συζητήσεις. Όσον αφορά τα ε, ζητήματα της εργασίας. Πρώτον, θέλουμε μια βαθιά συμφωνία. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κορμός της συμφωνίας θα πρέπει να εξετάζει και τις κοινωνικές πολιτικές. Ας σας δώσω κάποια παραδείγματα. Στις επενδύσεις, για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει ευθύνη των επενδυτών και αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τις συστάσεις του ΟΣΑ, τις συστάσεις του ΟΗΕ, τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά είναι συμφωνίες που θα πρέπει να αποτελέσουν τον κορμό της συμφωνίας στο κεφάλαιο της εργασίας. Δεύτερον, για τις υπηρεσίες. Όπως ανέφερα, θέλουμε να υπάρξει ένα ένας θετικός κατάλογος ε, δεσμεύσεων για να εξασφαλιστούν αυτές οι πολιτικές. Και πάνω απ' όλα, αυτό είναι σημαντικό για μας, όχι μόνο λόγω του αριθμού των ανθρώπων που εμπλέκονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες συμποσημειώσεις συμφωνίες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων. Και εκεί γίνεται αναφορά στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στις, διαπραγματεύσεις, ε, υποσημειώσεις, αλλά στο, σήμεν, στο, κύριο κείμενο, στο κύριο σώμα του κειμένου. Δημόσιες συμβάσει Και πάλι. Οι παρατηρήσει του ILO για τι συλλογικέ διαπραγματεύσει θα πρέπει να βρίσκονται στο κύριο κείμενο του κειμένου. Επίση, θα πρέπει να υπάρχει ρήτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Ο Ιγνάσιο αναφέρθηκε και στη γραφειοκρατία. Εμείς ε, θεωρούμε πιο σημαντικό τις, τις κόκκινες γραμμές μας, τις πολιτικές μας ε, αποφάσεις για, τα, για τους κανόνες εργασίας. Για το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως υπόθηκε, υπάρχει ήδη από ε, συμφωνίες. Δεν ξέρουμε αν ε, το μοντέλο των δύο πυλώνων είναι το σωστό, γιατί οι προθέσεις των Αμερικανών δεν είναι οι ιδανικότερες για μέσα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε είναι να υπάρχει ένα σύστημα που θα βελτιώνει διαρκώς και συστηματικά τους κανόνες εργασίας. Αυτό είναι ε, ένα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε είναι το γεγονός ότι οι ΙΠΑ δεν έχουν κυρώσει κάποιες από τις βασικές συμβάσεις που αναφερθήκαμε. Αλλά μιλάμε και για την εφαρμογή. Υπάρχουν και χώρες που έχουν κυρώσει αυτές τις συμβάσεις και στη συνέχεια δεν τις εφαρμόζουν. Δυστυχώς. Και νομίζω ότι σε αυτό μπορεί να συμφωνήσει αυτή η εμπορική συμφωνία. Άρα η εφαρμογή είναι Εξαιρετική σημασία. Στη συμφωνία με τον Καναδά αναφέρεται ότι θα καταβληθούν ε, οι προσπάθειες για να επικυρωθούν όλες οι συμβάσεις. Αλλά ε, δεν ε, υπήρχε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Με τσίπα είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να τις επικυρώσουν. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιοι άλλοι τρόποι εφαρμογής υπάρχουν. Ίσως θα μπορούσε ε, Ενδεχομένω να, να υπάρχουν άλλοι τρόποι με προστίκες ή προσαρτήματα στην ε, συνθήκη. Επίσης, όπως αναφέρθηκε στη συμφωνία με τον Καναδά, γίνεται αναφορά στις συμβάσεις πέραν και των βασικών συμβάσεων του κατευθυντών. Εμείς θέλουμε, εκτός από τις συμβάσεις του ILO, θέλουμε και κάποια από τα ευρωπαϊκά κοινωνικά πρότυπα να περιλαμβάνονται. Για τη δημοκρατία στο χώρο εργασίας, για παράδειγμα, που υπάρχουν σε κάποιες ευρωπαϊκές συμφωνίες, εμείς πιστεύουμε ότι αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο TTIP και επίσης κάτι τέτοιο θα πρέπει να ε, εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα. Δεν, χρειά, δεν είναι... Ε, δεν έχει νόημα να υπάρχει μια συμφωνία που θα ισχύει μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελών. Θα πρέπει και στο Τενεσί να μπορούν να πούνε. Επίση, θα πρέπει να ε, είναι υλοποιήσιμη η, η συμφωνία αυτή. Θα πρέπει να υπάρχουν απτέ κυρώσει και αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Οι διαπραγματεύσεις υπό τον ε, George Bush για παράδειγμα είχαν καταλήξει στο, σε συμφωνίες όπου υπήρχαν μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων. Δηλαδή λεγόταν ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις συγκεκριμένες. Και εμείς ενθαρρύνουμε και τους Αμερικανούς να το θέσουν αυτό ως ε, κόκκινη γραμμή. Τέλος, στο κεφάλαιο για την εργασία στην συμφωνία με τον ε, ε, Καναδά αναφέρεται η λέξη δεσμεύονται, δεσμεύσεις, αλλά δεν έχω λάβει σωστή απάντηση για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η δεσμευτικότητα που αναφέρεται εκεί. Και τέλος, θέλουμε έναν χρυσό κανόνα για τις ε, συνθήκες εργασίας. Η Επίτροπος μου είπε ότι θέλει μια να κάνουμε μια καινούρια αρχή, αλλά για να κάνουμε μια αρχή τέτοια θα πρέπει επιτέλους να ε, ε, επιλέξει ε, να σταματήσει αυτή η παράδοση της DigiTrade να μην θέλουν κυρώσεις. Σας ευχαριστούμε και τώρα κυρία Σάντος από την Business Europe. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα προσπαθήσω σήμερα να σας παρουσιάσω τη σκοπιά των εργοδοτών, αυτών που προσφέρουν τις θέσεις εργασίας. Νομίζω σημαντικό είναι να ξεκινήσω λέγοντας ότι ένα καλό επενδυτικό κλίμα, ένα καλό επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει καλές θέσεις εργασίας και η Business Europe και η ETUC ε, συζητούν εδώ και πολύ καιρό με κοινωνικούς εταίρους για να βεβαιωθούν ότι έχουμε το καλύτερο δυνατό μοντέλο για το εμπόριο ώστε να δημιουργηθούν στις θέσεις εργασίας και καλύτερες με καλύτερες αμοιβέ. Νομίζω από αυτήν την έννοια λοιπόν συμφωνούμε και οι δύο ότι χρειαζόμαστε καλύτερες και καλύτερα αμοιβόμενε θέσει εργασίας. Μια από τις προποθέσει για να έχουμε περισσότερες επενδύσει βεβαίως και στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπη. Και για να ε, επηρεαστούν οι Ευρωπαϊκέ Τρει Εργασία είναι να έχουμε μία μακροπρόθεσμη ατζέντα προτεραιοτήτων. Αυτό στην Business Europe για μα είναι πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε για το εσωτερικό ενδοευρωπαϊκό, μόνο κομμάτι. Πρέπει να υπάρξει νέα αγορά. Πολλά απομένουν σχετικά να γίνουν ακόμη στην Ευρώπη. Συζητήσαμε πολύ τι επενδύσει πρόσφατα και τι ε, συνθήκε και προποθέσει για να ξέρουμε ότι έχουμε βιώσιμη επενδυτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω. Πρέπει να αναφέρω και την ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και είναι ένα από τα σημεία όπου χάνουμε μεγάλους, πολλούς πόντους από την ανταγωνιστικότητά μας σε σχέση τουλάχιστον με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε σήμερα κάποιες εταιρείες, κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείες να εξαρτώνται από την ενέργεια. Να έχουν μια μεγάλη εξάρτηση από την ενέργεια, αλλά τότε ε, μεταφέρουν τις επενδύσεις τους προς τη ΣΥΠΑ γιατί το κόστος εκεί είναι χαμηλότερο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο ένα πλαίσιο που έχουμε ανάγκη νέων θέσεων και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, εκεί ανταγωνιζόμαστε με άλλες περιοχές εκτός Ευρώπης. Πολλές περιοχές στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ελκυστικότερες για τις επενδύσεις. Για μας λοιπόν η συμφωνία TTIP είναι και ένας τρόπος που εμείς ως επιχειρηματικός κόσμος πιστεύουμε είναι ένας τρόπος να δημιουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις για να γίνουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν θέσεις. Δεν θα μιλήσω για δεδομένα, δεν θα πω ε, τι γίνεται με τα ποσοστά απασχόληση. πόσες θέσεις θα δημιουργηθούν ή δεν θα δημιουργηθούν με τη συμφωνία TTIP. Όχι. Απλώς ένα θέλω να δηλώσω. Εφόσον υπάρξει συμφωνία και έχουμε μία ενιαία τοποθέτηση από τον επιχειρηματικό κόσμο, ε, που είμαστε θετικοί όλοι ταυτόχρονα. Η συμφωνία αυτή είναι η TTIP για την Κορέα. Όπως ξέρετε είχαμε τεράστιες συζητήσεις με την αυτοκινητοβιομηχανία, για την Ιαπωνία με άλλους συγκεκριμένους επαγγελματικού κλάδους. Στη συμφωνία TTIP σχεδόν όλοι από τον επιχειρηματικό κόσμο βλέπουμε να υπάρχει στήριξη και συμφωνούμε. Θεωρούμε ότι η συμφωνία θα είναι θετική για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και θα είναι πραγματικά θετική και για τι επενδύσει και για τις θέσει εργασία. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο τη βιωσιμότητα, και επειδή αυτό είναι μέρο των σημερινών μα συζητήσεων, καλωσορίζουμε την, ε, ε, τις εξελίξεις τις ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, όχι μόνο οι συμφωνίε έχουν εργατικέ και περιβαλλοντικέ ρήτρε. Αυτό είναι σχετικά νέα εξέλιξη. Όμω το αρχικό στάδιο ήταν όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ συμπεριέλαβαν τέτοιε ρήτρε στι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών και τώρα βλέπουμε αυτό να συμβαίνει και με περισσότερε αναπτυσσόμενε χώρε. Είναι θετική εξέλιξη όπως είπαμε, διότι μια εμπορική συμφωνία ουσιαστικά αφορά το εμπόριο, το να βελτιωθεί το εμπόριο ε, θέλει και το επενδυτικό κλίμα. Η κοινωνική και περιβαλλοντική συνιστόσα που είναι στον παρόδο είναι κάτι που προσπαθούμε να το συζητήσουμε. Το συζητάμε από το 1996 με την ατζέντα της Σιγκαπούρης αλλά ήταν, ε, ε, οι χώρες, ήταν λίγες οι χώρες τότε που ήταν έτοιμες να συζητήσουν ε, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνιστώσεις που επηρεάζουν το εμπόριο. Τώρα βλέπω να υπάρχει μάλλον καλή ε, πρόσληψη του όλου θέματος στο κοινό και να είναι όλοι πρόθυμοι να το συζητήσουν και στον ΠΟΕ ε, φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση και είναι ενδεχομένω η στιγμή να φέρουμε επιτάπητο τα δύο αυτά ζητήματα. Για μα, λοιπόν, στον επιχειρηματικό κλάδο πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο στοιχεία. Πρώτον, βεβαίω μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να περιλαμβάνει εργατικέ και περιβαλλοντικέ ε, ρήτρε και τα σχετικά κεφάλαια. Όμως αυτές οι διατάξεις δεν θέλουμε να είναι ένα είδος κρυφού ε, ανομολόγητο προστατευτισμού. Θέλουμε να υπάρχει παρόμοια προσέγγιση για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν αποκλήσει. Δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω χάρη την ίδια προσέγγιση στα ζητήματα αυτά. Μην πιστεύουμε λοιπόν και τρέφουμε την ψευδέστηση ότι θα έχουμε το ίδιο επίπεδο κοινωνικών ανησυχιών μέσω τη συμφωνία TTIP, ότι όλοι θα υποχρεωθούν σε αυτό. Εμεί ω Ευρωπαίοι, όπω ε, ανέφερε προηγουμένω και ο Τόμ, θέλουμε να εξάγουμε το κοινωνικό μα μοντέλο. Όμω πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το επίπεδο ανάπτυξη, να γνωρίζουμε ότι το επίπεδο ανάπτυξη σε πολλέ από τι χώρε με τι οποίε έχουμε διαπραγματεύσει δεν ισχύει αυτό για τι είπα βέβαια, αλλά στι άλλε χώρε μπορεί να μην είναι το ίδιο. Οπότε πρέπει να έχουμε υπόψη ότι όταν διαπραγματευόμαστε με μια χώρα όπω το Βιετνάμ, θα πρέπει να έχουμε διαφορετική προσέγγιση σε αυτού του είδου τα θέματα και όχι πράγμα που δεν συμβαίνει στις διαπραγματεύσεις μας με τις ΗΠΑ. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι χώρες θα πρέπει να εφαρμόζουν τη δική τους νομοθεσία. Σίγουρα να προοδεύσουν προς το σκοπό βελτίωσης της νομοθεσίας, αλλά σίγουρα με αυτονομία να εφαρμόζουν τα δικά τους, την εγχώρια νομοθεσία. Και κάτι που είναι μέρος μερικών εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την νομοθεσία ή να ε, αναθεωρούν την νομοθεσία για να προσελκύουν εμπόριο και επενδύσεις. Αυτό το πιστεύουμε και εμεί ακράδαντα. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο σύνολο προτύπων κοινωνικών και περιβαλλοντικών που δεν θα πρέπει να υποβαθμιστούν προκειμένου να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις ή να προωθήσουμε το εμπόριο. Ως προς το πεδίο τώρα. Ε, είναι σαφές ότι σήμερα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κυρώσει περισσότερες συμβάσεις ε, του ΑΕΛΟ, αλλά είδαμε ότι και στη συμφωνία με τον Καναδά, τη σφαιρική και σε βάθος ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, ε, περιλαμβάνονται ρήτρε για την αξιοπρεπή εργασία, κάτι που είναι καινούριο. Η συμφωνία λοιπόν αυτή έχει αυτό το καινοτόμο στοιχείο, θα πρέπει να το διατηρήσουμε και στη συμφωνία TTIP για τις δραστηριότητε CSR. Εδώ βλέπουμε για ε, κάποιες εταιρείες, ιδίως ευρωπαϊκές, για την εταιρική κοινωνική ευθύνη τα πράγματα είναι τελείω διαφορετικά. Το τι επίπεδο φιλοδοξιών έχουμε στην Ευρώπη κοινωνικό, σε κοινωνικά περιβαλλοντικά θέματα είναι ένα θέμα. Θα θέλαμε να γίνονται αυτά σεβαστά και εκτό Ευρώπη. Όμω δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ζούμε σε ένα κόσμο όπου δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα. Υπάρχει ένα ελάχιστο, ένα ελάχιστο νομικό πλαίσιο που δεν το καθορίζουν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε, το καθορίζουν τα κράτη, οι χώρε όπου εμεί ε, αναπτύσσουμε τι δραστηριότητέ μα. Δεν μπορούν λοιπόν οι εταιρείε, οι επιχειρήσει να αλλάξουν την υφιστάμενη νομοθεσία. Κάποιε φορέ Ό,τι μπορούμε να κάνουμε περιορίζεται, αυτά που μπορούμε να κάνουμε περιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχουν διατάξεις για την κοινωνική εταιρική ευθύνη, αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε μία μετριοπαθή προσέγγιση. Δεν ακολουθούν όλοι το ίδιο σύστημα με εμάς. υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα και πρέπει να είμαστε και βέβαιοι ότι συμμορφωνόμαστε με την ε, ε, υπάρχουσα νομοθεσία μιας χώρας. Αυτό αλλάζει πολύ με το αν έχουμε να κάνουμε με αναπτυσσόμενη ή ανεπτυγμένη χώρα. Επίσης πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι πρότυπα για τα εργασιακά και τα περιβαλλοντικά θέματα τις θέλουμε μεν, τα θέλουμε μεν, αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούν και να υλοποιηθούν. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό. Ο στόχος δεν είναι απλώς να περιλαμβάνονται διατάξεις, είναι να μπορούν να, γίνουν, να ε, εφαρμοστούν και στην πράξη. Το να έχουμε δεσμευτικές λοιπόν διατάξεις. Δεν εξασφαλίζει ότι θα ε, εφαρμοστούν. Είδαμε την περίπτωση της Γουατεμάλας, που είναι ένα παράδειγμα. Κάποιες φορές χρειάστηκαν έξι χρόνια για να φτάσει κανεί σε ένα σώμα διατησία. Με έναν επικοδομητικό λοιπόν διάλογο και με την ενεργό συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών, τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ καλύτερα. Μπορεί κανεί να πετύχει την ε, δραστική υλοποίηση. Οι κυρώσει, κατά την άποψή μα, δεν είναι λύση. Δεν είναι απάντηση αν θέλουμε βελτίωση των προτύπων σε όλε τι χώρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να αρχίσουμε το, τη συζήτηση. Ερωταπαντήσεις. Αλλά θα ξεκινήσουμε από το Προεδρείο. Με δύο-τρία λεπτά παρέμβαση για τον καθένα. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Κόνι Ρόιτερ και μετά ο κύριος Ραλφ Καμπχένερ. Ε, κύριε Ρόιτερ, έχετε το λόγο πρώτος. Προσωπείτε τη Σολιντάρη. Νομίζω με το κοινό των πολιτών, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε εστιάζει στα πρότυπα εμπορικά και απασχόληση. Και έχουμε τον κύριο Κάμπανερ εδώ. Στο Σιάτλ πριν από 7 χρόνια είχαμε συνεργαστεί. Όλοι επομένω ασχολούμαστε με αυτέ τι δραστηριότητε πολιτεία των πολιτών, τόσο ώστε να υπάρξει περισσότερη συνειδητοποίηση για ε, ε, αυτό το διακύβευμα. Άρα, καμπανάκι χτυπάει σήμερα το πρωί, γιατί είναι τόσο πρωί. Είναι το ότι δεν είναι περιπεπλεγμένη αυτή όλη η προβληματική για το TTIP και μιλώ ε, για το ότι θα πρέπει να ακούμε τους εμπειρογνώμενες για τους, ε, για τους δείκτες, για τα κριτήρια. Μόλις είναι έτοιμη συμφωνία προς υπογραφή για τα κοινωνικά πρότυπα μπορούμε να έχουμε αυτού του είδους τις διατάξεις για απασχόληση και έτσι να έχουμε ποιοτική απασχόληση. Γιατί μιλάμε για θέσεις απασχόληση, αλλά χρειαζόμαστε και αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι η καρδιά του Δήματος, να εξασφαλίσουμε οι συνθήκες εργασίας να είναι τέτοιες όπως τις θέλουμε και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Η διαδικασία να διαφορών θεωρούμε ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να υπάρχει κράτος δικαίου. Να μην έχουμε, να έχουμε μια ενιαία διαδικασία και όχι διαφορετική σε κάθε πλευρά του Ατλαντικού. Και ας κάνουμε αυτό το οποίο θεωρείται πιο δόκιμο πλευρά των επενδυτών. Το δεύτερο τώρα θέμα είναι κοινωνικές ε, διατάξεις του TTIP Μην έχουμε μίσουμε με τον Ομπάμα από τη μία και από την άλλη να υπομονωμεύεται το σύστημα αυτό το οποίο υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Να υπάρχει μία πολιτική κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, η προσέγγιση των θετικών σημείων. Είπαμε όχι αρνητική επαρρύθμιση. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μπορούμε να ξέρουμε και ποιες είναι οι θετικές εξελίξεις και όχι να λέμε τι αποκλείουμε και από την πίσω πόρτα να ξαναμπαίνουν τα προβλήματα. Όσον αφορά τώρα τον χάρτη της ε, αηφορίας, το σύστημα αυτό και με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας να έχουμε ε, άμεσα εφαρμόσιμα πρότυπα εργασίας. Επίσης, τα καλά νέα είναι ότι δεν έχουμε δύο διαφορετικού συνομιλητέ από Αμερική και από Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και από τι δύο πλευρέ, από τι δύο όχθε. Θα πρέπει τα Ευρωπαϊκά Όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν, να δείξουν ότι μπορούμε να έχουμε πρόοδο. Γιατί κάτι μπορούμε να καταφέρουμε. Άρα, πάρτε στα σοβαρά για τους φόβους και τους επικριτές και κοιτάξτε αυτά τα κριτήρια. Κοινωνική πρόοδος, ποιοτική απασχόληση και έτσι να υπάρχουν κοινωνικέ διατάξεις και νόμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. SME Europe. Ευχαριστώ κύριο Κάμπιονεν από την SME Europe. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Εκπροσωπώ την SME Europe, παρότι εργάζομαι για τη γυμνοκό μας. Η SME Europe είναι η συνομοσπονδία για τις ε, μικρομεσαίες Νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας έχουμε 20 εκατομμύρια τέτοιες επιχειρήσεις ε, που αντιστοιχούν στο 99% των επιχειρήσεων. Οι ΙΠΑ έχουν 38 τέτοιες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να ωφεληθούν και οι ίδιες και οι ε, εργαζόμενοι τους. Στα λίγα λεπτά λοιπόν που έχω στη διάθεσή μου θα ήθελα να επικεντρωθώ στην, ε, στις ε, διπλές, ε, στους διπλούς ελέγχους συμβατότητες που δημιουργούν πρόσθετο κόστος κατά μέσο όρο 20%. Στα καλλιτικά για παράδειγμα το κόστος αυτό είναι 35%. Στα, στην, στην φαντουργία είναι 20%. Στα τρόφιμα είναι πάνω από 50% και η έλεγχοι αυτοί αντιστοιχούν ως προς το κόστος τους σε δασμούς και έτσι η κατάσταση αυτή βεβαίως έχει αρνητικές επιπτώσεις και στα νοικοκυριά και στους καταναλωτές και μάλιστα υπήρχε και μια εκτίμηση από ένα ερευνητικό κέντρο της, Ευρώπης ότι κάθε νοικοκυριό θα μπορούσε να γλιτώσει 500 ευρώ κάθε χρόνο λόγω των ε, θετικών διατάξεων του TTIP. Για την απασχόληση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι γνωστές ως επιχειρήσεις που έχουν γενικά καλές σχέσεις με τους υπαλλήλους τους και στο πλαίσιο της σημερινής μας ε, συζήτησης θα ήθελα να πω ότι οι διατάξεις για, τις, ε, για τους ελάχιστους μισθούς, για τις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις που ισχύουν στην Ευρώπη δεν κινδυνεύουν ε, σε καμία περίπτωση από τις διαπραγματεύσεις για το TTIP. Αν σκεφτείτε μάλιστα τις δυνατότητες που μας ανοίγονται θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι μία από τις ευκαιρίες που έχουμε για την θέσπιση προτύπων διατλαντικών και είμαστε σε θετική θέση. Το TTIP λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Και θα ήθελα να σας καλέσω να δώσετε την ευκαιρία στις μικροβασίες επιχειρήσεις και στους υπαλλήλους σας να απολαύσουν τα ωφέλη του TTIP. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσατε πολλούς εμπειρογνώμονες και είναι πλέον η σειρά σας να θέσετε τα ερωτήματά σας. Αλλά σας παρακαλώ να είναι πολύ σύντομα και συγκεκριμένα τα ερωτήματά σας, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε την ευκαιρία να λάβουμε απαντήσεις από τους εμπειρογνώμονες. Δύο λεπτά θα πρότεινα, νομίζω ότι αρκούν. Η Μαρία Ρένα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να προλάβω πρώτα απ' όλα τρία θέματα επί της αρχής που έχουν λιγότερο να κάνουν με τα ζητήματα απασχόλησης. Πρώτον, το θέμα της επίλυσης διαφορών και κυρίως του επενδυτή κατά του κράτους, ISDS. Έχετε γνώση των αντιδράσεών μας σε σχέση με το θέμα αυτό. Τι δυνατότητα ρυθμιστική επιρροή θα υπάρχει εδώ και κυρίω προ τα θέματα τη απασχόληση. Έπεισα το φόρουμ τη ρυθμιστική συνεργασία. Είπατε ότι σήμερα πρέπει να απαλλαγούμε από τους διπλούς ελέγχους ε, κατά κύριο λόγο και αναφέρατε το θέμα των ε, φαρμάκων, της χημία και από την άλλη, είπατε και για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Εγώ δεν ξέρω πολλέ ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει που να λειτουργούν σε αυτό το τομέα και να είναι θύματα των διπλών ελέγχων. Νομίζω λοιπόν το ρυθμιστικό πλαίσιο που λέτε είναι ψέμα ότι θα ευνοήσει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και έπειτα για τον αρνητικό κατάλογο που αναφέρθηκε προηγουμένω. Είτε είναι πρωτοβουλία είτε αρνητικό κατάλογο, καλό θα ήταν να υπάρχει η εγγύηση ότι εφόσον θελήσουμε μπορούμε να επανέλθουμε σε άλλη νομοθεσία προ το γενικό συμφέρον των Ευρωπαίων. Σε γενικέ λοιπόν γραμμέ αναφερθήκατε και νομίζω ότι ο καθένα εδώ είτε από την πλευρά τη εργοδοσία είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφερθήκατε σε μελέτε αντικτύπου που μα φαίνονται υπερβολικά φιλόδοξε. Πώ λαμβάνετε υπόψη τι μελέτε αντικτύπου, που είναι πολύ αριθμε σήμερα και είναι λιγότερο αισιόδοξε από τι δικέ σα. Θα έλεγα μάλλον απεσιόδοξε. Λόγου χάρη έχουμε τι αναλύσει των ε, συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που έχουν γίνει ε, εδώ και μία δεκαετία και βλέπουμε ότι υπήρχε μια συμφωνία που προέβλεπε τη δημιουργία ενό εκατομμυρίου θέσεων εργασίας ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε και τελικά υπάρχουν λιγότερες 600.000 θέσεις περίπου. Και επίσης ε, βλέπουμε ότι η κοινωνική προστασία στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν ήταν πολύ ψηλή υποβαθμίστηκε. Αυτό επηρέασε ε, ίσως την αγοραστική δύναμη των Μεξικανών γιατί η συμφωνία ήταν μεταξύ ΙΠΑ και Μεξικού. Όχι. Η αγοραστική δύναμη των Μεξικανών μειώθηκε 7 φορές. Δηλαδή η πρόσβαση στα αγαθά των Μεξικανών αυξήθηκε κατά 2,5 7. Βλέπουμε ε, σήμερα ότι συμφωνίε όπω αυτή ε, αποδεικνύουν ότι δυσκολίε υπάρχουν. Δεν είμαστε κατά των συμφωνιών. Αλλά δώστε μα επιχειρήματα που θα μα επέτρεπαν να ε, σκεφτούμε συμφωνίε που δεν είναι όπω αυτή η συμφωνία του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών. ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα. Αφενός τα εργατικά πρότυπα. Η δεν είναι απλά μια χώρα που δεν έχουν εγκρίνει κάποιες από τις συμβάσεις του ILO, αλλά που παραβιάζουν τις συμβάσεις αυτές. Στο Τενεσί πρόσφατα έγινε προσπάθεια να απαγορευτεί η ίδρυση Συμβουλίου Εργαζομένων σε εργοστάσιο της Volkswagen. Οπότε πώς ακριβώς ε, θα διαμορφωθούν οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών, τι μορφή θα έχουν, θα ε, ε, εξασφαλίζονται δικαιώματα συνδικαλιστικά. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι το ζήτημα των θετικών επιπτώσεων. Οι θετικές επιπτώσεις λόγω του, με, της αύξησης του εμπορίου υπάρχουν ε, οικονομικά ωφέλη. Όταν όμως ε, ε, θα πρέπει να, όμως να υπάρξει και διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι τομείς και περιφέρειες θα υποστούν διαφορετικού χαρακτήρα επιπτώσεις. Οπότε το ερώτημα είναι ποιοι τομείς θα ωφεληθούν ποιες περιοχές και περιφέρειες θα ωφεληθούν, ποιοι τομείς και ποιες περιοχές θα χάσουν και πώς ακριβώς θα αντισταθμιστούν αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις σε, αυτές τις, ε, σε αυτούς τους τομείς και σε αυτές τις περιφέρειες γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια ανισομετρία στην Ευρώπη όσον αφορά την ανάπτυξη υπάρχουν αξιολογήσεις, έχουν γίνει μελέτες από την πλευρά της Κομισιόν για να αξιολογηθεί αυτό το ζήτημα και αν ε, όχι αν έχει δώσει ε, εντολή η Κομισιόν να γίνονται τις μελέτες και αν όχι γιατί όχι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιατσουβίτσια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να, ευχαρισ... να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις σας. Ήταν πολύτιμες προτού καταλήξουμε σε αποφάσεις ή προτού ξεκινήσουμε σοβαρά να εργαζόμαστε επί του TTIP. Ορισμένοι μας επέστησαν την προσοχή ότι οι διατάξεις θα πρέπει να είναι υλοποιήσιμες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να το προσέξουμε γιατί στο χαρτί μπορεί κανείς να καταγράψει διάφορες, ε, διάφορους κανόνες αλλά αν πρακτικά δεν είναι εφαρμόσιμοι κανόνες ε, αυτοί τότε δεν έχει νόημα να τους θεσπίζει κανείς. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξής. Μπορείτε να μας πείτε ποια, ποια είναι τα βασικά πρότυπα εργασίας που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην συμφωνία αυτή. Να μας τις κατανομάσετε. Και μια ερώτηση για τον εκπρόσωπο των Ευρωπαϊκών ε, Συνδικάτων. Είπατε ορισμένα πράγματα για την αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Το ερώτημά μου προς εσάς είναι το εξής. Ποιο εργαλείο θα πρέπει να συμπεριληφθεί ώστε οι επιχειρηματίες να έχουν κίνητρο να δημιουργήσουν ασφαλείς θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες για τις συνεισφορές του σήμερα το πρωί. Βλέπω ότι υπάρχει μια ποικιλία απόψεων και οπτικών γωνιών. Είναι σημαντικό αυτό για να ξέρουμε πώς προχωρούν οι διπλωματεύσεις. Η γενική μου εντύπωση είναι ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που θα απαντηθούν, διότι δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει ίσως να υπάρχει ένα πρώτο κείμενο, σχέδιο συμφωνίας πριν μπορέσουμε να κάνουμε συγκεκριμένα σχόλια. Επίσης, καλωσορίζω την άποψη του SME Europe που είπε ότι για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας μπορεί να είναι ενδεχομένως πολύ θετική η εξέλιξη από τη συμφωνία TTIP και για τις επιχειρήσεις και για το επενδυτικό κλίμα και για το ISDS να πω ότι το θέμα δεν είναι βασικά το κράτος δικαίου το οποίο θα συνεχίσει να υπάρχει. Το θέμα είναι αν μπορούμε να προσφέρουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους για να επενδύσουν στην Ευρώπη. Ε, ε μπορούμε να τους κάνουμε να είναι ασφαλείς για επενδύσεις στην Ευρώπη όπως έχουμε πει τόσες φορές και έχουμε δει να συμβαίνει και από την άλλη πλευρά της μάχης. Αλλά για την ε, διάσταση των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών θεμάτων ε, στην ε, συμφωνία. Κύριε Μπερσέρο, ήθελα να μου πείτε, εάν θα υπάρξουν όντως, ε, αν θα υπάρξει όντως ενδελέχης και εξέταση των κεφαλαίων αυτών στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε, η κυρία Κάρη. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες για αυτές τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους. Μόλις συναντήθηκα με δανούς πυροσβέστες και τους εκπροσώπους τους και μου είπαν ότι έχουν τεράστια προβλήματα στο εργασιακό τους περιβάλλον, διότι υπάρχουν ε, επικίνδυνες χημικές ουσίες και πρωτεσίλες το, η συμφωνία TTIP ήδη δημιουργεί πολλά προβλήματα για αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο και βεβαίω είναι σημαντικό το εργασιακό του περιβάλλον. Εάν θέλουμε να έχουμε κοινού κανόνε, πώ μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε του ίδιου κανόνε, αλλά ταυτόχρονα θα προστατεύουμε του εργαζομένου και θα έχουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Πώς αυτά τα δύο δεν θα αντιφάσκουν μεταξύ τους. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε τις επιπτώσεις στην απασχόληση που θα προκύψουν από τη συμφωνία TTIP. Αλλά μιλάμε για 600.000 θέσεις με 1.200.000 θα περάσουν σε εμείς πολιτήσεις. Ισχύει αυτό. Κυρία Βάρνα, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ε, για τις δημόσιες προμήθειες, είναι το ερώτημά μου. και εμείς δεν θεωρούμε ότι ο αρνητικός κατάλογος είναι κατάλληλο εργαλείο για τη διασφάλιση των δημόσιων υπηρεσιών. Το αντίθετο, είναι μια εξέλιξη που πρέπει να την αποτρέψουμε. Σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, οι αποτυχημένες ιδιωτικοποιήσεις έχουν αποδείξει πόσο αρνητικές επιπτώσεις είχαν στις, στα εργασιακά δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις για το TTIP βρίσκονται σε εξέλιξη και οι διαπραγματεύσεις για το TISA, για το Trade and Service Agreement, και έχουμε άλλη μια φορά μια πλήρη απελευθέρωση ή μια κίνηση προς την πλήρη απελευθέρωση των υπηρεσιών και μάλιστα ανεπρίσ, ανεπίστρεπτα. Ε, αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτή την ε, συμφωνία ότι ό,τι ιδιωτικοποιηθεί άπαξ δεν θα επιτρέπεται να κοινωνικοποιηθεί ποτέ ξανά. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την ύπαρξη των πολιτών στην Ευρώπη και γι' αυτόν τον λόγο σας ρωτάω, ιδιαίτερα εσάς κύριε εκπρόσωπο της Κομισιόν, μπορείτε να μας εξασφαλίσετε σήμερα, εδώ και τώρα, ότι ούτε το TTIP ούτε το TISA θα ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση για ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων ε, προμηθειών και ότι στους τομείς αυτούς θα εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη και να γίνονται σεβαστά τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπαλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ερώτηση. Η μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν λέει το όνομα του τι θα γίνει με την ε, απασχόληση γιατί σήμερα. Μήπως έχουμε μια συγκριτική μελέτη όσον αφορά το τι έχει γίνει στο παρελθόν σαν μελέτε όσον αφορά τις ελεύθερες συναλλαγές. Έχουμε δηλαδή κάποιο είδους ε, σημαντική έρευνα όσον αφορά τις προηγούμενες προβλέψεις ακριβώς ε, όπως είπε η συνάδελφος η παρακαθήμενη πριν από λίγο δεύτερον. Κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω. Εάν σήμερα δεν έχουμε κάποιο περιορισμό στο ρόλο του γραφείου εργασίας, τι απάντηση θα δοθεί σε σχέση με ένα πρότυπο ευρωπαϊκό στο οποίο θα, πάμε και όχι ένα αμερικανικό. Αν μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτό το στοιχείο. Τρίτο, θεωρητικά τι γίνεται στον πρώτο ανταγωνισμό για τις ε, ε επενδύσεις. Σταθερή η ελεύθερη διακίνηση, θέλουμε ελεύθερη κυκλοφορία και μήπως έτσι καταλήξουμε σε κάποιο είδους μείωση της αμοιβή της εργασίας. Γιατί βλέπουμε συνέχεια τέτοιο φαινόμενο σήμερα. Τη Συμφωνία Ελληνά με ναύτα. Άρα μήπως τελικά φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Κάτι άλλο. Εμείς οι σοσιαλιστές είμαστε κατά το ότι δηλαδή το TTP τι θα γίνει αν έχουμε μια πολυεθνική η οποία μπορεί να προσφύγει δικαστικά κατά κάποιο κράτος όσον αφορά το, την κοινωνική νομοθεσία για το ISDS. Σας ευχαριστώ. Δύο θέματα έχω να θέσω. Για την απασχόληση. Τι είναι για εκεί που περιμένουμε να υπάρξει ε, αύξηση τη θέση απασχόληση σε κάποιες περιφέρειες γιατί δύο των τους ε, μας είπαν ο καθένας τελείως διαφορετικά πράγματα για το κατά πόσο δεν θα έχουμε περισσότερες ή λιγότερες θέσεις απασχόλησης. Οπότε και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπεσέρο πρώτα. Πώς Πώ σχολιάζε αυτά που είπε ο κύριο Τζένγκιν, πώ θα ήταν πιο σωστό να έχει περισσότερε εισβάθου μελέτε η λιγοτερε θεσει απασχοληση οποτε και εγω θα ηθελα να ρωτησω τον κυριο μπεσέρα πρωτα πω σχολιαζει αυτα που ειπε ο κυριο τζεγκιν πως θα ηταν πιο σωστο να εχει περισσοτερε ει βαθο μελετες η ευρωπαικη επιτροπη οσον αφορα την απώλεια θέσεων απασχόλησης Είναι πολύ αυτό το θέμα. Μήπως το που μας οδηγεί, λέτε, σε καλύτερη απασχόληση ή όχι. Όσο τώρα όσον αφορά τα πρότυπα της απασχόλησης. Πριν ακούσαμε τον πρέσβευτη τον κύριο Γκάρνερ και μας είπε δεν μπορούν είπα να εγγυηθούν την εφαρμογή των προτύπων του ΑΕΛΟ. Αλλά θα συμμορφωθούν. Αυτό σηκώνει συζήτηση. Κύριο Τζένκινς μας είπε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το TTIP αντί της κύρωσης των ε, ε προτύπων απασχόληση από τη ΣΥΠΑ. Προσπαθώ να καταλάβω πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Και τι θα γίνει με την κύρωση. Και επίσης τελευταία μου ερώτηση προς τον κύριο Μπεσέρα. Γιατί δεν έχει συζητηθεί το κεφάλαιο για την απασχόληση καθόλου. δεν είναι αυτό Στι συνομιλίε με τη ΣΥΠΑ μια προτεραιότητα. Ευχαριστώ Αγνούς, ο Σούλτσε. Αξιότιμο κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ε, συζήτηση αυτή, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν χαίρομαι καθόλου για το γεγονός ότι ακούστηκαν πάρα πολλά ε, αρνητικά πράγματα ο κατάλογος των αρνητικών στοιχείων για το TTIP είναι πολύ μεγαλύτερος από τα θετικά που ακούστηκαν και είμαι σίγουρος ότι αν η συζήτηση κινηθεί μόνο γύρω από τα αρνητικά δεν πρόκειται να, να στεφτεί με επιτυχία το TTIP. Μιλάμε διαρκώς για τη δημιουργία νέων θέσεων ε, απασχόλησης και υπάρχει και μια... ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα ε, ε, προβλέψει τις περισσότερες ε, ε, θέσεις εργασίας. Μήπως θα πρέπει να συζητήσουμε πόσες ε, θέσεις απασχόλησης όμως θα χαθούν αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για το TTIP. Δεν είναι προτιμότερο περισσότερο να υπάρχουν ε, οι θέσεις απασχόλησης και να τις διατηρήσουμε εδώ από το να έρθουμε μετά από 15-20 χρόνια και να ε, διαπιστώσουμε ότι οι θέσεις απασχόλησης χάθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ασία. Η συζήτηση λοιπόν ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί στα θετικά και όχι μόνο στα αρνητικά. Λοιπόν, έχω 7 ακόμη ομιλητές στον κατάλογο ομιλητών μου. Ο κύριος Κέλλερ. Έχω ένα απλό ερώτημα. Γνωρίζουμε ότι η συμφωνία αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΙΠΑ έχει ως σκοπό να καταργήσει τους μη δασμολογικούς ε, φραγμούς. Μας διαβεβαιώνουν διαρκώς ότι δεν θα μειώσει τα πρότυπα, την, την προστασία των εργαζομένων, στην υγεία, στην ασφάλεια, αυτή η συμφωνία. Πώς μπορεί η συμφωνία να βελτιώσει όμως ε, όλα αυτά. Η συμφωνία με τον Καναδά ε, περιλαμβάνει περισσότερες από χίλιες ε, σελίδες και οι σελίδες που είναι αφιερωμένες στα, εργατικά δικαιώματα είναι μόλις πέντε. Όλοι αναφέρουν τα τεχνικά, τις τεχνικές προδιαγραφές για τις αυτοκινητές βιομηχανίας Αυτός θα είναι ο τρόπος, λοιπόν, θέλετε να μας πείτε, που θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ η κυρία Λόπες Φερμιέρο. Σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε. Πρώτα-πρώτα, μερικοί από εσά επιμένετε να θεωρείτε ότι αυτή η συμφωνία είναι πάρα πολύ καλή για την ε, απασχόληση. Όμως, σε σχέση με τη συμφωνία ναύτα, οι Αμερικάνοι εργαζόμενοι ξέρουν ότι χάθηκαν τότε ένα εκατομμύριο ιδέε Ευρωπαίοι εργαζόμενοι, ξέρουν ότι οι εγγυήσει δεν αρκούν και ότι πρόκειται να έχουμε χαμήλωμα του πύχη για τα πρότυπα τα εργατικά. Τι γίνεται με αυτά τα οικονομικά μοντέλα τα οποία ελαχιστοποιούν την ε, ζήτηση, ιδίω σε, σε μη ανταγωνιστικού. Βρισκόμαστε τώρα σε φάση αντιπληθωρισμού. Και σε άλλους τομείς έχουμε τώρα πάρα πολλέ απολύσεις. Και γνωρίζετε ότι μια που δεν έχουμε δημοκρατικά όργανα που να επιτρέπουν τη μόνιμη αναθεώρηση της συνθήκης από όταν υπογραφηθεί και ούτε έχουμε ε, συνδικάτα διατλαντικά ούτως υπήν, τότε λίγες είναι αυτές οι που έχουμε όσον αφορά αυτό, τα, τα δίκτυα παραγωγής και επενδύσεων που είναι πολυεθνικού χαρακτήρα. Επίσης, μας λέτε ότι θα υπάρξει αναγνώριση των εργασιακών δικαιωμάτων από τη ΣΥΠΑ. Επίσης έχουμε και ένα σωρό συμφωνίες του Γραφείου Εργασίας για επιθεωρήσεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις κλπ. Και έχουμε και τις ενημερωμένες συνθήκες που όμως δεν έχουν κυρωθεί. Θα γίνει και αυτοί οι κύρωση και αν θέλουν να κυρώσουν γιατί δεν προσυπέραψαν τόσες συμφωνίες. Και τι θα γίνει με τις ρήτρε και τα εργατικά θέματα όταν δεν έχουν καν κυρώσει τις σχετικές συμφωνίες η Αμερικανία. Ο κύριος Μαρίν. Ναι, Μαρίν, Μαρίν, Μαρίν. Ça doit être Monsieur Εννοείται ο κύριος Μαρτά. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, εγώ ήθελα να σταθώ σε μια φράση, τέλο πάντων δύο λόγια, που μα είπε ο εκπρόσωπο τη Business Europe όταν τάχθηκε υπέρ ενό διαλόγου με, με του εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών για την επίλυση των διαφορών. Με εκπλήσει, διότι σε αυτή τη συμφωνία οι συνδικαλιστικέ οργανώσει και το Ευρωκοινοβούλιο έχουν αποκλειστεί πλήρω από κάθε γνώση για τι διαπραγματεύσει, για το άνοιγμα των κεφαλαίων. Με εκπλήσει λοιπόν αυτό που αναφέρατε. Και ε, επιπλέον, ε, πρόσφατα, συναντήσαμε την αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει αναλάβει ίδια τι διαπραγματεύσει. και ε, αναγνώρισαν, παραδέχτηκαν οι ίδιοι ότι στην συμφωνία αυτή θα υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Η πραγματική ερώτηση είναι ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι και ποιοι χαμένοι τελικά. Ποιοι θα είναι οι χαμένοι, μιλάμε για την απασχόληση αλλά μιλάμε και για μοντέλα, έτσι. Μιλάμε για το ευρωπαϊκό ε, μοντέλο έναντι του αμερικανικού. Αυτό που συμβαίνει στι Ηνωμένε με τη διαχείριση των υδάτων λόγω χάρη και όπου τι Αμερικανικέ ε, πόλει τις ε, έχουν ε, πλήξει οι πολυεθνικές και μάλιστα με δικαστικές αποφάσεις γιατί απλώς επερασπίζονται τα γενικό συμφέρον τι μπορείτε να μα διαβεβαιώσετε εσεί ότι θα γίνει με το νερό εδώ. Μπορείτε να μα δώσετε ένα παράδειγμα Διεθνού Συμφωνία με του Αμερικανούς που δεν επέβαλαν εκείνη το δικό του το μοντέλο στου άλλου. Αυτό είναι ακριβώ ο κίνδυνο. Το ευρωπαϊκό μοντέλο θα καταρρεύσει ε, στην, από την πίεση του Αμερικανικού. Οι θέσει εργασία θα αρχίσουν να φεύγουν από εδώ και από εκεί. Και θα ε, σταματήσουμε ω Ευρώπη να είμαστε οι μεγάλη μεγάλοι και να επιβάλλουμε του δικού μα περιβαλλοντικού εργασιακού και κοινωνικούς Ευχαριστούμε κυρία Μάκεντάιρ. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ανησυχώ για το γεγονός ότι ο ρόλος της Επιτροπής Απασχόλησης δεν θα πρέπει να είναι μόνο η προστασία των εργαζομένων, όσο σημαντικό και αν είναι αυτό το θέμα, αλλά και το ζήτημα της ε, δημιουργίας ε, νέων θέσεων εργασίας. Και χάρηκα που άκουσα για τι 20 εκατομμύρια ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε ότι το 85% των θέσεων απασχόληση δημιουργούνται από μικρός, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε ο σκοπός του TTIP είναι προφανώς να απελευθερωθούν οι εμπορικές συναλλαγές και οι επενδύσεις, να καταργηθούν ε, φραγμοί, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά και σε υπηρεσίες. Δηλαδή να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να σας πω ότι ε, ανησυχώ για το γεγονό ότι οι πολίτες μας ε, παραπληροφορούνται. Λαμβάνω εκατοντάδες email που μου λένε ότι θε, επίκειται ψηφοφορία για, τη, για το TTIP. Εδώ δεν έχουμε καν κείμενο. Οι διαπραγματεύσεις από το κείμενο θα ξεκινήσουν του χρόνου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να διακρίνουμε τους μύθους από την πραγματικότητα και οι συζητήσεις μας θα πρέπει να βασίζονται στην πραγματικότητα και όχι σε κάποιους συναισθηματισμούς και κάποιες ανησυχίες οι οποίες μπορεί και να βασίζονται σε λάθος δεδομένα. Για παράδειγμα, εγώ ε, είμαι ευγνώμων ε, σε οργανώσεις όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη στην Βρετανία που εξέδωσε έγγραφο για, την, για το διαχωρισμό μεταξύ μύθου και πραγματικότητας που δεν εκδόθηκε δηλαδή από πολιτικούς αλλά εκ μέρους ενός οργανισμού που ξέρω ότι έχει προβληματισμούς γιατί ακούγονται και ιδέες ότι το, το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας δεν θα είναι αναγνωρίσιμο και αυτό δεν ισχύει οπότε θέλω να ακούσω από τους ειδικού στο πάνελ πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό ακριβώ, να διακρίνουμε τους μύθου από την πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πολύ. Το απλό ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου είναι ποια είναι τα ωφέλη Θέλουμε να μας πείτε κύριε Μπερσέρο ποια, είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα ωφέλη και σε ποια βάση δεδομένων ε, έχετε κάνει τις προβλέψεις σας. Και αυτό που μας αφορά είναι και η ποιότητα των θέσεων εργασίας. Δεν θέλουμε καταρτισμένους ανθρώπους να τους μετατρέψουμε σε μη καταρτισμένους, αλλά θέλουμε να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για το μέλλον της Ευρώπης. Για την εκπρόσωπο του ILO Είμαι θετικά διακείμενη γενικά ως άνθρωπος ε, και θα ήθελα να μου πείτε κάποια θετικά παραδείγματα συμφωνιών όπου συμπεριλαμβάνονται ή όπου ε, ενισχύθηκαν τα πρότυπα συμμετοχής των εργαζομένων και όχι απλά να, ερχόμαστε και να λέμε ότι τι ωραία καταφέραμε και ε, εξασφαλίσαμε τα πρότυπά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Μινόε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τα όσα είπε η κυρία Κόλλη Κολυμπάλη και εγώ δεν είμαι βέβαιη ότι η συμφωνία TTIP θα βοηθήσει πάρα πολύ τους εργαζομένους μου φαίνεται ότι μάλλον θα αρχίσουν να τρέχουν ε, πανικόβλητοι με όσα πρόκειται να συμβούν. Θα είναι κάτι σαν ολοκαύτωμα. Επίσης ακούσαμε και την Business Europe να μας λέει ότι δεν περιμένει να υπάρξουν σοβαρές αλλαγές ως προς τα εργασιακά δικαιώματα. Ο κύριος Τζένκινς συμφωνεί ότι υπάρχει μια σειρά από ριζικές αλλαγές που πρόκειται να έρθουν προς το μέρος μας, αλλά ότι θα τις αντιμετωπίσουμε και λέει ότι δεν θα υπάρξουν σοβαροί τριγμοί. Ξέρει όμως μάλλον πόσες δουλειές χάθηκαν σε ανάλογες περιπτώσεις διεθνών συμφωνιών και επίσης θα ξέρει και τι έγινε με τη Συμφωνία Ναύτα στις ΗΠΑ. Πολιτείες. Μπορώ να στείλω και στη συνάδελφο Ιονγκέριους αν τα θέλει. Εσείς λοιπόν μπορείτε να πείτε ότι δεν θα υπάρξουν απώλειες στις τέσσερις εργασίες και ότι οι εργασιακές εξελίξεις θα είναι θετικές. Ευχαριστούμε. Ναι, ναι, οι εξαγωγές, όπως είπα, χρειάζονται πάρα πολύ τη σημερινή μέρα. Όμως, το θέμα είναι θα υπάρξουν περισσότερες θέσεις απασχόλησης, περισσότερο εμπόριο, αλλά χρειάζονται και κοινέ διαδικασίες, ε, κοινά πρότυπα. Τι γίνεται μέσα με το TTP, πώς θα προσεγγίσουν οι αγορές. Για τον Γιώργο Καμπιόνερ, ερώτηση. Το ISDS με τις ΜΜΕ. Τελευταία στοιχεία που άκουσα είναι ότι μία υπόθεση κόστησε από 8 έως 30 εκατομμύρια δολάρια. Οι επιχειρήσεις που εκπρόσωποι θα ωφεληθούν Τι θα γίνει, ποιος θα πληρώσει την ύφη, το κράτος οι διαπραγματευτέ μπορούν να μα πούν τι θα βγει από το ISDS. Κύριε Χάρκιν. Ευχαριστούμε του προσκεκλημένου μας για όλε τι απόψει που μα εξήγησαν και πριν σα ρωτήσω να σα πω ότι είμαι από κάποια χώρα. Την Ιρλανδία που έχει ρυθμού ανάπτυξη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα σήμερα στην Ευρώπη. Και αυτό γιατί έχουμε ζωντανό πολύ εμπόριο με τη ΣΥΠΑ. Οι ερωτήσει μου είναι οι εξή. Μάλλον επικριτικού χαρακτήρα. Άκουσα να δει συναδέλφοι ότι ίσω ε, ε, οι συμφωνίε αυτέ θα βοηθήσουν το εμπόριο, αλλά θέλω να ρωτήσω πρώτα-πρώτα την Επιτροπή. Με αυτό το πρότυπο αξιολόγηση απασχόληση που έχετε, μήπω υπάρχουν και άλλα τέτοια μοντέλα, γιατί η θεωρητική σας βάση οδηγεί σε Πολύ πολύ σημαντικέ επιπτώσει σε σχέση με τα στοιχεία στο οποίο καταλήγεται. Και λέμε για δημιουργία πολλών θέσεων απασχόληση, αλλά για να δούμε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ. Η ανεργία είναι χαμηλή. Όμως ε, εμείς εδώ είμαστε μάλλον στάσιμη σε επιδόσεις μας. Θα πρέπει να εξορροπήσουμε τα πράγματα και να έχουμε ως στόχο και την ποσότητα και την ποιότητα. Κυρία Κόλλη, από το Γραφείο Εργασίας είπατε ότι ένα από τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι το πώς θα είμαστε συνεπείς με τις διατάξεις που διέπουν το Γραφείο Εργασίας. Έχετε κάποιο πρόγραμμα από τώρα μπορείτε να το ξεκινήσετε τόσο ώστε να εξασφαλίσετε αυτή την συνέπεια για το πλέγμα διατάξεων του ΑΕΛΟ. Και τελευταία ερώτηση προς τον κύριο Τζέκινς από τη Συνομοσπονδία. Είπατε κάτι για κόκκινη γραμμή. Of τι γίνεται με τη συμφωνία με τον Καναδά. Για εφισταμένη συμφωνία μπορούμε να επικαλεστούμε το ISDS. Μήπως εκ των υστέρων μπορούμε να μπαλώσουμε τα πράγματα, δηλαδή όσο δεν πάνε καλά με αυτή τη συμφωνία. Και ο ίδιος ο Γιούνκερ το είπε επίσης ότι Δεν είναι και τόσο ε, απαραίτητο το SDS, μια που ήδη έχουμε συστήματα απονομή δικαιοσύνη ε, άρτια. Πώς επηρεάζει το SDS τι διαφωνητεύσεις. Ω προ Ως προς τις δυνατότητες του TTIP να παράσχει έναν χρυσό κανόνο κανόνα για την εργασία και το περιβάλλον. Μου κάνει πάντοτε εντύπωση και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Όταν ακούγεται ότι, όταν αναφέρεται ότι η συμφωνία με τον Καναδά είναι ένας χρυσός κανόνας, ένα καλό πρότυπο για την βιώσιμη ανάπτυξη, το ΣΥΤΑ, αν το εξετάσατε, αυτή η συμφωνία με τον Καναδά είναι πιο κάτω και από την ΝΑΦΤΑ και ε, περιλαμβάνει χαμηλότερα πρότυπο όσον αφορά την ε, η ναύτα περιλαμβάνει και κάποιες διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια. Το, η συμφωνία με τον Καναδά σε καμία περίπτωση δεν το κάνει αυτό. Οπότε ανησυχώ πραγματικά. Χρησιμοποιούμε την ΣΥΤΑ ε, ως μοντέλο για το TTIP. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε υπομοσπονδιακό επίπεδο όσον αφορά τα δικαιώματα συνδικαλιστικής οργάνωσης, συλλογική διαπραγμάτευσης. Οπότε από αυτή την άποψη ε, ένας χρυσός κανόνας για ε, τα εργατικά δικαιώματα. Μάλλον θα πρέπει να είναι ε, ένας συνδυασμός των καλύτερων πτυχών και από τις δύο πλευρές. Και τέλος, για τις επενδύσεις. Το ανέφερε ο Τόμ πολύ σύντομα, αλλά υπήρχε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αφορά το κεφάλαιο για την προστασία των επενδύσεων. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ότι το κοινό θα έχει εμπιστοσύνη στο ότι θα προστατεύονται οι επενδύσεις του, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχα κριτήρια συμπεριλαμβανομένων και των ε, γραμμών του ΟΕΣΑ. Μήπως τελικά ε, το TTIP είναι μια ευκαιρία για να δημιουργηθούν ε, κανόνες σε αυτό το τομέα. Επίσης, ευχαριστώ η κυρία Λάμπερτ δεν είχαμε δει το, την κάρτα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να επανέλθω στην κοινωνική συνιστόσα, διότι είμαστε και στην Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ξέρουμε ότι οι υγειονομικέ υπηρεσίε και οι κοινωνικέ υπηρεσίε είναι από τι πιο σημαντικέ περιοχέ απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μα θέλουμε να μείνει έτσι και για το μέλλον. Και βεβαίω είναι ένα τομέα που ενδιαφέρει ιδιαίτερω το κοινό και εμά. Και βεβαίω μπορούμε να συγκρίνουμε τα πράγματα με το τι έγινε στη συμφωνία με τον Καναδά, την ε, ε οικονομική και εμπορική συμφωνία και να δούμε ποιο είναι το ύψος των ε, φιλοδοξιών μας. Να δούμε τι έγινε με τις δημόσιες προμήθειες, την πρόσβαση στην αγορά. Πιστεύω ότι στην απελευθέρωση κανείς μπορεί να προχωρήσει μόνο και όχι να οπισθοδρομήσει. Οπότε, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τόσο μεγάλες δυσκολίες προκειμένου να ορίσει τα τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντας, συμφέροντος συγγνώμη, στις δικές μας τις ίδιες τις οδηγίες και επειδή δεν είναι σαφές αν υπάρχει διάταξη για το μονοπόλιο της προσφοράς υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου εξηγήσει διότι οι υπηρεσίες αυτές απλώς δεν εξαιρούνται από τις διαπραγματεύσεις TTIP. Οι διαβεβαιώσεις που έχουμε τώρα όταν κοιτάζουμε τους ορισμούς είναι ότι οι υπηρεσίες που ακούμε δεν καλύπτονται επαρκώς ε, από τους ορισμούς που ήδη έχετε συντάξει. Πιστεύω ότι θα ανακοφίζονταν πάρα πολύ δημόσια γνώμη αν απλώς εξαιρούσατε αυτό ε, το κομμάτι. Ή τέλος πάντων να υπήρχε ένας ορισμός που να ξεκαθαρίζει ότι οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος ε, είναι εκτός και οι υπηρεσίε κοινωνική, οι εταιρείε κοινωνική πρόνοια, δημοσίου συμφέροντο, ανησυχούν για το τι επιπτώσεις θα υπάρξουν για αυτέ από τη συμφωνία. Θα χρειαστούμε λοιπόν σαφεί ορισμού. Ευχαριστούμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στου εμπειρογνώμονέ μα με την αντίστροφη σειρά. Θα δώσω το, ρόλο το λόγο στο Ραλφ για κάποιε συγκεκριμένε απαντήσει. Παρακαλώ σύντομα και με ταχύτητα. Ευχαριστώ κύριε Λάγκε για την ερώτηση της κυρίας ε, Νάτι. πάντοτε σεβόμαστε την διμερή κανότητα των κρατών να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συμβάσεις. Αυτές συμπληρώνουν την ευρωπαϊκή πολιτική και προσφέρουν επιπλέον προστασία στους επενδυτές που ιδάλλως δεν θα μπορούσαν να προσφύγουν κατά των κρατών. Ήδη από τη δεκαετία του 50 οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ξεπεράσει τις 1500 διμερείς ε, συμφωνίες πέραν των 400 συμφωνιών που προβλέπονται. Οι ε, συμφωνίες λοιπόν αυτές ουσιαστικά καθησυχάζουν τους επενδυτές που χρειάζονται εμπιστοσύνη, νομική βεβαιότητα και ασφάλεια. Και όλες αυτές οι συνθήκες συμβάλλουν στον ίδιο σκοπό. Βλέπω λοιπόν το ίδιο πλαίσιο να διαμορφώνεται και εδώ και νομίζω ότι θα είχε νόημα να το δούμε και η αυτή τη σκοπιά για τις διαπραγματεύσεις TTIP. Έπειτα, ακούγοντα τα όσα συζητήθηκαν εδώ σήμερα, έχω την εντύπωση ότι Προσπαθούμε να δούμε τι δημοτεύσει τύπου από την άποψη τη ανάπτυξη και των θέσεων εργασία που μα απασχολούν γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για το 2020 όμω και του στόχου του, μιλάμε για την ε, παγκοσμιοποίηση των ευρωπαϊκών επιχειρησιών, πώ μπορούμε μέσω τη ευρωπαϊκή πολιτική να προσφέρουμε ανάπτυξη και θέσει εργασία στου πολίτε. Είναι ευκαιρία για τον δημοσιοτομέα η συμφωνία TTIP. Ε, Δεν υπάρχουν δύο συστήματα, ένα ευρωπαϊκό και ένα ε, αμερικανικό. Υπάρχουν σφάλματα σε όλα τα... και στις δύο υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευθούν τα, τα δικαιώματα ε, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κράτη, σε πολιτείες της, των Μιλάμε για τις θέσεις εργασίας, αλλά σκεφτήκαμε την ε, ποιότητα και το σε ποιους τομείς δημιουργούν. Υπάρχει μια αναφορά που συχνά την ξεχνάμε. Δεν μιλάμε μόνο για βιομηχανικές σχέσεις εργασίας. Μιλάμε... Ο σημαντικότερος τομέας αυτή τη στιγμή είναι η υγεία. Ο μεγαλύτερος εργοδότης στη Γερμανία είναι η Κάριτας και όχι η Volkswagen. Και η κοινωνική οικονομία απασχολεί το 12% του εργατικού δυναμικού. Οπότε δεν θέλουμε να υπονομευθούν οι διατάξεις ε, για αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν εμπόδια που έχουμε ε, ξεπεράσει. Θέλουμε να μιλήσουμε για την ποιότητα των ε, υπηρεσιών, για την ποιότητα της απασχόλησης. Αυτό είναι το βασικό. Και να πω ότι δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τις υπάρχει ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας και υπάρχουν μεγάλες επενδύσεις που ξεκινάν από την Ιρλανδία και στη συνέχεια περνούν στις ΗΠΑ και είναι ένας μηχανισμός που έχει αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστος Οπότε αυτό πρέπει να το ε, καθορίσουμε. Η υγεία δεν είναι αντικείμενο εμπορίου. Σάντο. Ρωτήθηκε το ρόλο των συνδικάτων της κοινωνία των πολιτών. Θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε τις συμβουλευτικέ και υποπτικέ ομάδες για την Κορέα. Λειτουργεί το σύστημα. Πολλά βέβαια μπορούν να βελτιωθούν. Και σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει να παρακολουθήσουν το κεφάλαιο εφορία. Όλοι εμπλέκονται. Και οι οργανώσει της κοινωνία των πολιτών. Όσον αφορά τη συμμετοχή της κοινωνίας και των συνδικάτων για τις διαπραγματεύσεις. Δεν θα υπησταθώ σε λεπτομέρειες, αλλά όλοι γνωρίζετε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε διαφάνεια. Όλοι συμμετέχουμε εκεί και νομίζω ότι υπάρχει συμμετοχή και τάση για περισσότερη συμμετοχή. Έχουμε συζητήσει πολλά για την ποιότητα των θέσεων απασχόληση για τις επιπτώσεις της Συμφωνίας Ναύτα. Για μην ξεχνάμε ότι μιλούμε για εταίρους σε διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης. Μεξικό, Καναδάς, ΗΠΑ. Όταν μιλάμε για ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούμε για δύο εταίρους με παρόμοια ανάπτυξη. Ένα αυτό. Το άλλο είναι ότι η ναύτα συνήθω πάνω από 20 χρόνια πριν. Θα μιλούμε για νέα συμφωνία σε νέο πλαίσιο με διαφορετικούς κανόνες, νέους κανόνες. Ελπίζω ότι κάτι έχουμε διδαχθεί. Άρα από μια συμφωνία σε διαφορετικό πλαίσιο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε πρότυπο του παρελθόντος. για το μέλλον. Μπορούμε να συζητήσουμε τι είδους θέσεις απασχόλησης θα ε, έχουμε. Αλλά όπως προείπα, δεν θέλω τώρα να πούμε συζήτηση για αριθμητικά στοιχεία. Παναβάνω πρώτη για μια συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ κλάδων της οικονομίας. Αυτά σε επαναλαμβάνω από όσα είπα στην εισήγηση. Τζέγγινς. Γιατί δεν είμαστε κατά της TTIP. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει πάντως. Είμαστε κατά της ΣΕΤ. Πάμε ότι έχουμε τις κοινές γραμμές, έχουμε το ISDS, προστασία κρατικών υπηρεσιών και επίσης να έχουμε εφαρμογή των ε, τάξεων απασχόλησης. Δεν πειράζει για όλα αυτά το ότι Ο είπε ο Ιγνάσιο, όπως είπαμε για την απασχόληση. Αυτό είναι template και για το SDS είπαμε ότι είναι άλλο σύστημα ανακύπτει και για το ΣΕΤΑ και για το TTIP Επομένως εδώ έχουμε θέμα συνέπειας ότι γίνεται στην μια και τη λέμε στην άλλη αλλά δεν φταίμε εμείς γι' αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στήριζονται στο εμπόριο Όμως, πέρα από το τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις, είναι το θέμα πολιτικό για το τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι πολιτικό, όχι οικονομικό. Άρα, θέλουμε ψηλά πρότυπα. Να, παράδειγμα, για τα προϊόντα της χημικής βιομηχανίας, αν το δεχτούν οι Αμερικανοί, που δεν νομίζω, κάτι σαν το REACH, αν το δεχθούν, και αν έχουμε τα πρότυπα του REACH διατλαντικά, φανταστικό. Να, και θα πρέπει να κάνει ο υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει να εφαρμόσει σχετικά πρότυπα το πριν από χρόνια για τι νανοτεχνολογίε. Αν εκεί έχουμε ψηλά πρότυπα για τέτοια ζητήματα, καλώ. Αλλά δεν θέλουμε να κατεβάσουμε τον πύχη με τι διαπραγματεύσει. Και το Διεθνέ Γραφείο Εργασία, χωρί να μπούμε στι λεπτομέρειε, έχουμε 8 πρότυπα για συλλογικέ συμβάσει εργασία, για εργασία ανηλίκων ε, και ε, εργασία, που αποφύγη διακρίσεων. Έχουμε την ε, διακήρυξη του 98 και όλα τα μέλη του Γραφείου Εργασία θα πρέπει να τα εφαρμόζουν όλα αυτά και φαντάζομαι μπορεί θα περισσότερα έχει πρόσωπο του γραφείου. Και μας είπαν και άλλο. Έχω εδώ ολόκληρη λίστα με τέτοια πρότυπα του ΆΕΛΟ Αυτά θεσπίστηκαν όταν ήταν ο Μάντελσον στην Γενική Διεύθυνση τη Απασχόληση. Άρα Καταλαβαίνετε πόσο παλιά είναι. Τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Εμείς θεωρούμε ότι ισχύει ό,τι λέμε εμείς. Έχουμε σύστημα λήψη αποφάσεων δημοκρατικό. Δεν, δεν τα βάζω το κεφάλι με αυτά που σας λέω. Υπάρχει διαφορά μεταξύ διαφάνειας και επικοινωνίας. Πολλοί σε Συμβουλίο και Κομισιόν ενδιαφέρονται περισσότερο για επικοινωνία παρά για διαφάνεια. Και η επικοινωνία δεν είναι πάντοτε ένα πραγματικό περιστατικό. Είχαμε την τελευταία τριμερή τη κορυφής για κοινωνικές υποθέσεις και τι είπε για τη συμφωνία με την Κορέα ο Μπαρόσο. Όλα πολύ καλά πάνε είπε. Δεν ισχύει αυτό όμως, δεν είπε την αλήθεια. Δεν θα πρέπει να το ξέρω και δεν υπάρχει αιστείας. Τι είναι αυτό το πράγμα, το περιστατικό, είναι θέμα ε, διαφήμισης και επικοινωνία. Και και εμάς πρέπει καλά τα πάει, όμως είπε και εκείνη ότι είναι στο DNA της η διαφάνεια. Και την άλλη μέρα είπε ένα δημοσιογράφο στην Ιαπωνία, μπορεί να δούμε τα έγγραφα για την συμφωνία Ιαπωνία Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όχι, λέγε τόση διαφάνεια, του είπε την άλλη μέρα. Να, είδατε τι γίνεται με το DNA και τη διαφάνεια. Uh, Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο λόγος στην κυρία Κόλλη Κουλαμπαλή. Πολλές ερωτήσεις προς τον ΑΕΛΟ. Ευχαριστώ να είναι πολλές ερωτήσεις προς τον ΑΕΛΟ, προς την, ε, εφαρ... την κύρωση από τις ΗΠΑ, 8 ε, συμβάσεων του ΑΕΛΟ. Όντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ε, έχει κάποια αντίρρηση με, τις, με τους μηχανισμούς παρακολούθησης του ΑΕΛΟ και έχει συμπληθεί και στην ε, βασική δήλωση όλων των μέλων του ΑΕΛΟ πόλη έχω να προσπογράψω του 98. Τώρα για τα υπόλοιπα σχόλια, πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα πρότυπα και να επηρεάσουμε τις εμπορικές συμφωνίες με τα εργαλεία που έχουμε από τον ΑΕΛΟ. Αυτό το κάνουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε με τις προτεραιότητες για την εξωπρεπή εργασία. Εκεί υπάρχει συνοχή με τα όσα κάνει ο ΑΕΛΟ, διότι υπάρχουν οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις του ΑΕΛΟ που επηρεάζουν τα τέσσερα βασικά πρότυπα για την εργασία που έχουν να κάνουν με τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Εκεί που υπάρχουν ε, ελλείμματα στην, ε, στα εργασιακά δικαιώματα και όπου κάποια χώρα έχει κάτι να κάνει σε τομεακό επίπεδο και σε μικρό επίπεδο για ακριβώ τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Αυτά, αυτά καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν στην εμπορική συμφωνία, ώστε ζητήματα που έχουν συγκεκριμένε ευαισθησίε για έναν τομέα, για την βελτίωση πρώτη σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, να καλυφθούν. Νομίζω η εμπορική συμφωνία ανοίγει και την πόρτα σε μηχανισμούς συνεργασίας. Ε, ναι, γιατί έχουμε μια συμφωνία μεταξύ ανεπτυγμένων χωρών, οπότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις βελτιστές πρακτικές των ΜΕΝ και των ΔΕ με μηχανισμούς που θα επιτρέψουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με καλύτερο διάλογο των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και τη γενικότερη αναβάθμιση των προτύπων. Τώρα, για το τι είναι φήμη και τι πραγματικότητα. Ε, μια μελέτη αντικτύπου που έχει γίνει εξάντε είναι μύθος κατά τη δική μου άποψη, διότι Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ υποθετικά τα πορίσματα. Ένα επιπλέον τρόπο θα ήταν να υπάρχουν συστηματικέ εξάντια αναλύσει για να στηρίζουν τι μελέτε αντικτύπου και να βλέπει κανεί και εκ των υστέρων ποιο ήταν ο αντίκτυπο, ώστε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που, τυχώς, που τυχόν ε, προκύπτουν. Αυτό θα προέβλεπε, θα επέτρεπε μια πολύ αυστηρότερη παρακολούθηση και υλοποίηση των ε, ε, διατάξεων. Δόθηκαν κάποια παραδείγματα για περιπτώσεις όπου τα πρότυπα βελτιώθηκαν. Εγώ ανέφερα τουλάχιστον τρία τέτοια στην παρουσίασή μου ήταν τα παραδείγματα που εμείς εξεύγαμε στη μελέτη μας και είχαν να κάνουν με την αιρεσιμότητα πρώτης κύρωσης, δηλαδή εκεί όπου οι χώρες πρέβλεψαν νομοθεσία για να βελτιώσουν το ρυθμιστικό και νομοθετικό τους πλαίσιο ε, για τα εργασιακά πρότυπα και ως συνέπεια της εμπορικής συμφωνίας. Αυτός, αυτό συνέβη τουλάχιστον ε, στη συμφωνία ΝΑΦΤΑ με το Μεξικό. Αλλά είδαμε και αλλού ε, να συμβαίνει κάτι με την συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Καμπότζης. Διαβάστε τη μελέτη και θα τα και ως προς την συνοχή. Ναι, υπάρχει συνοχή μεταξύ των εργαλείων του ΑΕΛΟ, πιστεύουμε εμείς, αλλά ένα από τα πράγματα που προσπάθησα να αναπτύξω στην παρουσίασή μου ως προς την συνοχή για τις εμπορικές συμφωνίες είναι ότι δεν μπορούμε μόνο να ξεχωρίζουμε και να απομονώνουμε κάποια εργαλεία του ILO με πολύ ε, περίεργη και περίπλοκη γλώσσα που κάνει πολύ δύσκολη την εφαρμογή των προτύπων. Το να συμπεριλάβουμε κάτι στην εμπορική συμφωνία απλώς γιατί ακούγεται ωραίο. Μπορεί να δυσχεράνει πάρα πολύ ε, το τι θα κάνει κανείς μετά και προσπαθώντας συμβουλευτικά και διοργανωτικά να δει πώς θα τα ε, υλοποιήσει και να δει κατά πόσον υπάρχουν παραβιάσεις στη συνέχεια ή όχι. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντική συμβουλή. Και τώρα η Ιγνάσιο. Ευχαριστώ πολύ. Απευθύνθηκαν κάποια ερωτήματα σε μένα, οπότε με συγχωρείτε αν δεν καταφέρω να απαντήσω σε όλα. Θα προσπαθήσω όμως να απαντήσω σε όσο περισσότερα ερωτήματα γίνεται. Θα προσπαθήσω να δομήσω τις απαντήσεις μου σε τέσσερις κατηγορίες. Οφέλη του TTIP, κίνδυνοι, μελέτες και το ζήτημα του κεφαλαίου εργασίας. Να ξεκαθαρίσω όμως το εξής. Πρόκειται για μια διαπραγμάτευση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ ισότιμων μερών η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να έχει κανένα κόμπλεξ στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Δεν πρόκειται για μια διαπραγμάτευση όπου οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν τα δικά τους πρότυπα σε εμά. Ούτε το αντίστροφο. Η συμφωνία αυτή θα βασίζεται στην ισορροπία στις αξίες των ε, δύο μερών και εκεί όπου υπάρχουν ε, κάποιες διαφορές, γιατί υπάρχουν διαφορετικές ε, κοινωνικά πρότυπα στις δύο πλευρές, αυτές οι διαφορές θα παραμείνουν. Αλλά κοιτάμε να διαπραγματευτούμε σε εκείνους τομείς όπου οι αρχές μας είναι κοινέ. Εκεί που υπάρχουν διαφορές ενδεχομένως να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη ρυθμιστική συμβατότητα αλλά η συμφωνία αυτή δεν έχει σκοπό σε καμία περίπτωση τη μείωση του επίπεδου προστασίας μας. Είτε, αφορά αυτό την, είτε μιλάμε για την εργασία είτε για το περιβάλλον. Θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρά κεφάλαια και για τα δύο αυτά θέματα και σε καμία περίπτωση δεν θα υπαναχωρήσουμε από τις δικές μας αρχές και τις δικές μας αξίες προστασίες. Κάποιοι σας εκφράσατε σκεπτικισμό όσον αφορά τις, τους ισχυρισμού ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να ωφελήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή να δημιουργήσει ωφέλη στο ρυθμιστικό τομέα. Ε, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά να σας πω κάποια παραδείγματα. Αν ε, έχεις μια μικρομεσαία επιχείρηση που ε, παράγει στην Ευρώπη ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή γενώσιμα φάρμακα, για να κάνεις εξαγωγές της ΕΠΑ, θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να υποβληθούν σε έλεγχο του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων της, ε, των ΙΠΑ ακόμη και αν έχεις λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλεις να εξάγεις βελγικά μήλα στις ΙΠΑ πρέπει να περάσει από μια πολύ περίπλοκη ε, γραφειοκρατική διαδικασία 6-7 ετών ορισμένες φορές προκειμένου να πάρεις άδεια για να κάνεις εξαγωγές. Αυτό, ε, αυτά τα στοιχεία του ρυθμιστικού καθεστώτο μας ε, δεν έχουν καμία σχέση με την ε, προστασία. Απλά αυτό που δεν έχει, ε, σε αυτό στο οποίο δεν έχει δοθεί σημασία είναι πώς μπορούν να, να ε, καταργηθούν εμπόδια μέχρι τώρα. Και συζητούμε και για τα χημικά προϊόντα υπάρχουν κάποιοι τομεί όπου μπορεί κανείς να αποφύγει περιττές υποβολές εκθέσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ε, αποδυναμώσουμε την εφαρμογή του κανονισμού REACH. Κάποιοι θα το ήθελαν, αλλά Όπω ακριβώ εμείς δεν πρόκειται να αλλάξουμε τα πρότυπά μας, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε και το αντίστοιχο στις ΗΠΑ. Αν δει κανεί λοιπόν τον τομέα τη μεταποίηση, θα δει ότι μέσω της κατάργησης των ε, δασμών και μέσω της κατάργησης τη επικάλυψης των ελέγχων, ενδεχομένω, μπορεί να δημιουργηθεί ένας τομέα ε, λειτουργικός, για την εξαγωγή μεταποιημένων προϊόντων από και προς ε, τις ΕΠΑ, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ δηλαδή. Ποιοι είναι οι τομείς όπου φοβάστε ότι θα αμφισβητήσουμε ε, το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης. Δημόσιες υπηρεσίες. Σαφέστατος θέλω να είμαι δεν έχουμε αναλάβει καμία δέσμευση όσον αφορά την απελευθέρωση οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας. Έχουμε, ανεξάρτητα από το αν θα είναι ε, αρνητικός κατάλογος, υπάρχει η δημοκρατική αρχή ότι αν Ακόμη και αν ε, κάποιο τομέα έχει ιδιωτικοποιηθεί, έχει απελευθερωθεί, μπορεί στο μέλλον να επανακοινωνικοποιηθεί. Να είμαι σαφή. δηλαδή δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τι δημόσιες υπηρεσίε, Ξέρω ότι πολλοί στο συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχουν πιστεί αυτό και φυσικά με χαρά μου θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή, αλλά μπορώ να σα βεβαιώσω ότι δεν αμφισβητείται το δικαίωμα μελλοντικών κυβερνήσεων να προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες κοινωνικές, στέγασης για παράδειγμα. Αν κάτι τέτοιο θα πρέπει να θεωρεί, θα θεωρεί η κυβέρνηση αυτή ότι θα πρέπει να παρέχει τη δημόσια, τότε αυτό θα εξασφαλίζεται. Επίσης, οι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες προμήθειες στην Ευρώπη ε, χωρίς κανέναν ε, περιορισμό. Αυτό δεν ισχύει όμως για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στις ΕΠΑ. Ποια είναι η ανησυχία λοιπόν που έχει εκφράσει, έχουν εκφράσει κάποιοι στο συνδικαλιστικό κίνημα και στην Επιτροπή σας εδώ ξέρω ότι υπήρχαν πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις όσον αφορά την ε, οδηγία για τις ε, δημόσιες προμήθειες και υπάρχει πλέον διάταξη ότι θα πρέπει να ε, οι αρχές δημόσιων προμηθειών και συμβάσεων θα πρέπει να εφαρμόζουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Το κείμενο που έχουμε αυτή τη στιγμή και το οποίο συζητούμε με τις ΕΙΠΑ έχει βελτιωθεί όσον αφορά την, τις δημόσιες ε, συμβάσεις με βάση τις δικές μας οδηγίες. Για το ερώτημα για το ISDS δεν μπορώ να κάνω μια μεγάλη παρουσίαση για το θέμα αυτό διότι η Κομισιόν πολύ σύντομα θα δημοσιεύσει μια έκθεση των ε, έπειτα από τις διαβουλεύσεις Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχω εξουσιοδότηση να μιλήσω για το θέμα αυτό, για το SDS, δεν μπορώ να το κάνω σήμερα, αλλά με χαρά μου να έρθω κάποια άλλη στιγμή, σε κάποια άλλη περίσταση, κάποια άλλη συζήτηση. Για το ζήτημα των μελετών. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε σχέση με τις δυνατότητες του TTIP. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή ε, είναι υποθετικές ε, γιατί δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για την οργάνωση και υπάρχουν πάρα πολλές ε, μεταβλητές. Οι περισσότερες μελέτες προβλέπουν ωφέλη που συνάδουν και με την μελέτη επιπτώσεων που είχε υποβάλει και η Κομισιόν. 0,5% αύξηση του ε, ΑΕΠ σε 10 χρόνια προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλες οι επιπτώσεις στην οικονομία. Όχι, σε 10 χρόνια θα είναι 0,5% η αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό θα γίνει, όχι αυτό που ακούστηκε στη συζήτηση ότι θα διαρρέσουμε αυτό το 0,5% δια 10 χρόνια. Δεν συμβαίνει αυτό. Προκειμένου να ε, εκτιμήσεις μια κατάσταση θα πρέπει να λάβεις υπόψη όλους τους ε, παράγοντες και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,5% μετά από 10 χρόνια. Αλλά πάντοτε προσέχαμε στις μελέτες μας να μην συμπεριλάβουμε συγκεκριμένο αριθμό για το ε, ε, απασχόλησης που θα δημιουργηθούν γιατί ε, δεν μπορεί να, να γίνει μια σαφής πρόβλεψη για αυτό το στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι τα δεδομένα μας δείχνουν ότι 5 εκατομμύρια ε, θέσεις εργασίας στην Ευρώπη εξαρτώνται από το εμπόριο με τις υπακιά, και αν οι εμπορικές συναλλαγές αυξηθούν λόγω της συμφωνίας, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση των θέσεων εργασίας. Πόσες θα είναι αυτές, δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Και αυτός είναι ο λόγος που θα συμφωνήσω ότι δεν θα πρέπει μόνο να κάνουμε μελέτες για το μέλλον, αλλά να αξιολογούμε και συμφωνίες ε, που έχουν ήδη γίνει. Όπως είπε και η Λίσα, υπάρχουν ε, διαφορές μεταξύ των ε, συνθήκων είπα και Μεξικό, αλλά οι διαφορές αυτές είναι πολύ διαφορετικές που υπά... από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να δούμε μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την... και το ελεύθερο εμπόριο. Είδατε Έχετε υπόψη σα την ε, συμφωνία με την Νότια Κορέα. Όταν το συζητήσαμε εκείνο το θέμα, εδώ στο Κοινοβούλιο υπήρξαν πάρα πολλέ ερωτήσει όσον αφορά τι επιπτώσει που θα είχε στην ευρωπαϊκή ε, μεταποίηση στο, ως προς το γεγονός ότι υπήρχε πολύ μεγάλο έλλειμμα της Κορέας σε σχέση με, στο εμπορικό της ισοζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι οι επιπτώσεις λοιπόν αυτής της συμφωνίας. Υπάρχει τεράστια αύξηση εξαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κορέα για πολλούς λόγους, όχι μόνο για την ε, εξαιτία της ε, συμφωνίας. Αλλά είναι ένα παράδειγμα συμφωνίας που έχει επιφέρει θετικές, ε, θετικά αποτελέσματα για την Ευρώπη και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε δεδομένο, ως δεδομένο ότι δεν θα είμαστε σε θέση ε, να ε, καταλήξουμε σε μια ε, παρόμοια συμφωνία με τις ΗΠΑ. Δύο-τρία λόγια για τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν λέμε ότι αυτό που κάναμε στη συμφωνία με τον Καναδά είναι και ακριβώς το δείγμα για το τι θα πρέπει να επιδιώξουμε στη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Προσπαθούμε απλώς να πάρουμε τα δύο σύνολα των καλύτερων στοιχείων και από τις δύο προσεγγίσεις. Ε, πρέπει να απλουστεύσουμε τα πράγματα όπως την υλοποίηση όπως είπατε, διότι ότι έχουμε και στη συμφωνία με τον Καναδά και με την Κορέα είναι, δεσμευτικ... είναι δεσμευτικές ρυθμίσεις για την εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα έπειτα για την διατησία με το ανεξάρτητο σώμα μεσολαβητών δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της συμφωνίας. Απλώς τα εμπορικά ζητήματα δεν μπορούν να γίνουν θέμα επιβολής που εξαρτάται πάρα πολύ από την κοινή γνώμη. Δηλαδή αυτό που ισχύει είναι ότι όποτε υπάρξουν προσφυγές για εργασιακά υπερβαλλοντικά λαμβάνουν μεγάλη προβολή στο κοινό. Ό,τι συμβεί σε σχέση με αυτά τα πρότυπα γνωστοποιείται πολύ γρήγορα στο κοινό και πιέζει πάρα πολύ την κάθε χώρα. Οι ΙΠΑ όντως έχουν δεχτεί εμπορικέ κυρώσεις που δέποτε εφαρμόστηκαν στην πράξη. Τώρα έχουν περάσει μόλις τη φάση της ε, εκδίκασης, αλλά οι διαφορές για εργασιακά δικαιώματα στις ΙΠΑ ε, φιλτράρονται και μόνο εάν αποδειχθεί ότι υπήρξε παραβίαση των βασικών αρχών του ΑΕΛΟ και υπήρξε κινητικό αντίκτυπο για το εμπόριο, μόνον εφόσον αυτό τεκμηριωθεί, τότε μόνον η υπόθεση μπορεί να περάσει στο μηχανισμό επίλυση διαφορών. Αυτό δεν ισχύει στη δική μα την προσέγγιση. Στη δική μα την προσέγγιση, εφόσον υπήρξε ε, παραβίαση των βασικών αρχών του ΑΕΛΟ, αυτό επιτρέπει την ε, προσφυγή και την εκδίκαση υπόθεση ασχέτω με το τι επίδραση υπήρξε στο εμπόριο ή όχι. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό τη Κορέα. Έχουμε και οι δύο συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών με την Κορέα και εμείς και είπα με ένα κεφάλαιο για τα εργασιακά. Στην Κορέα δεν είχαν επαρκή δικαιώματα και δικαίωμα έκφραση στο δημόσιο τομέα τα, συνδικαλιστικές οργανώσεις. Εμείς το συζητήσαμε με την Κορέα για την υλοποίηση της συμφωνίας, αλλά είναι λίγο δύσκολο να θυμίσουμε να επηρεάσουμε το τι θα γίνει στην περίπτωση των ΗΠΑ και των δημοματεύσεων μα μαζί του εδώ, διότι εκεί θα πρέπει να αποδειχθεί επιπλέον και ο αρνητικό αντίκτυπο για το εμπόριο. Είναι λοιπόν περίπλοκη συζήτηση, αλλά σίγουρα πρέπει να αναζητήσουμε μια θετική προσέγγιση. Απλώ να προσθέσω τα πράγματα λέγοντα ότι οι συμφωνίε των ΗΠΑ τι δίνονται να εφαρμοστούν, οι ευρωπαϊκέ όχι. Ο πρόεδρο, δύο πλέον ερωτήσει. για το κεφάλαιο, για την απασχόληση. Είπαμε για τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Πώς αντιδρά στην πρότασή μας για την κάλυψη των εργασιακών ε, το κράτος των ΗΠΑ. Επίσης, είπατε ότι τώρα ετοιμάζεται μια πρόταση για κεφάλαιο για την αηφορία. Ποιος το κάνει αυτό. Αν έχω δίκιο, υπάρχει μια συμβουλευτική ομάδα που θα πρέπει να συμβουλεύσει την Επιτροπή. Και το Γραφείο Εργασία επίσης, εάν του ζητηθεί. Αλλά και το Κοινοβούλιο έχει κάποια εμπειρία Συζητιέται μαζί με όλα αυτά τα συμβολιστικά ε, σώματα το θέμα ή όχι. Ε, Α, είναι και μια άλλη ερώτηση που πρέπει να σας απαντήσω τώρα. Η ερώτηση που μου υπέβαλαν ότι δεν ε, δίνουμε αρκετή προτεραιότητα όσον αφορά. Αυτή την πλευρά Πρώτα-πρώτα. Είναι σωστό αυτό που είπατε έχουν υποβάλει αυτό το εντέλεχε σύγγραφο Τα σχετικά με την αγορά ανάπτυξη. Για την πλευρά της απασχόλησης και του περιβάλλοντος. Τα συζητήσαμε με τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες, λεπτομερή σχόλια και μας εξήγησαν τι κάνουν για αυτούς τους δύο τομείς. Ακόμα πάντως δεν έχουν ε, αντιπροτείνει κάτι. Ίσως για τα θέματα θα είναι τόσο επίμαχα όσον αφορά τις ε, διαταντικές διαπραγματεύσεις. Uh, in the context of the Trans-Pacific uh, negotiations. Να δούμε πώς θα προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις. Και να δούμε πώς θα δημορφωθούν οι προτάσεις μας και η Γενική Διεύθυνση για το κλίμα, για το περιβάλλον, για την απασχόληση και, για το εμπόριο. Όλοι, όλοι. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ήρθαμε σε επαφή και με, το, με την ε, ομάδα της, της συμβουλευτική και όταν η πρόταση έχει ολοκληρωθεί, τότε θα την κοινοποιήσουμε και στα κράτη-μέλη. Και με την ε, ομάδα παρακολούθησης της ε, ΙΝΤΑ, της Διεθνής για το Εμπόριο, και κοινοποιούμενα όλα αυτά στα κρατημέλη, τότε θα δημοσιοποιηθούν. Όποιος θέλει μπορεί να τα μελετήσει. Ε, δεν θα είναι μόνο η ΣΥΤΑ, θα έχουμε και άλλα στοιχεία. Θα βελτιώσουμε αυτά που κάναμε στην ΣΥΤΑ. Ευχαριστώ να ακούσουμε τις ε, παρατηρήσεις σας. Και δεν συμφωνώ με, τον με κύριο Ντάλιν που είπε ότι ε, είναι λιγότερο δεσμευτική μία συμφωνία από την άλλη, από την ίδια συμφωνία δηλαδή με την Κορέα. Είσαι πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για ερωτήσεις και για απαντήσεις. Πάρα πολύ δύσκολο να συνοψίσει κανείς όλα αυτά που συζητήσαμε. Το ένα θέμα είναι η συνέχιση τη απασχόληση, το άλλο είναι οι κρατικέ υπηρεσίε, οι δημόσιε υπηρεσίε. Επίση το άλλο θέμα, το καλό θα έχουμε θέσει απασχόληση. Το τέταρτο επίση μεγάλο ερώτημα είναι τι είδου θέσει απασχόληση θα είναι αυτέ, εάν υπάρξουν. Αυτά είναι τα ερωτήματα στο οποίο θα πρέπει να επανέλθουμε. Και με εσά και με κύριε Μπεζέρο και με τους υπόλοιπους ε, εμπειρογνώμονες. Αυτή ήταν μόνο η πρώτη ακρόαση για την απασχόληση, αλλά σίγουρα θα πρέπει να επανέλθουμε. Και σίγουρα θα δουλέψουμε πολύ εντατικά για αυτά τα θέματα και για τη συμφωνία TTIP. Ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να ακούσετε τις ε, ερωτήσεις και να μας ε, απαντήσετε με όλα αυτά τα στοιχεία που έχετε. Με τις ερωτήσεις τώρα μπορείτε να προσμεστείτε περαιτέρω και να επανέλθετε σε λίγους μήνες. Και σας ξανά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.